Dear friends, dear colleagues, we would like to start the session because we have very limited time for... Ας αρχίσουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για τους ε, προσκεκλημένους μας. Οπότε ας ε, σας ευχηθώ καλώς ορίσατε αρχίζοντας την συνεδρίαση και σας ε, ενημερώνω ότι πρόκειται για την συνέχιση της πρωινής συνεδριάσεως που συζητήσαμε για τα δικαιώματα για την ελεύθερη διακίνηση, για ζητήματα συνεργασίας αστικού δικαίου και θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε την δημοκρατική διάσταση σε σχέση με τις ε, ευρωπαϊκές εκλογές την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και επίσης θα πρέπει να καθορίσουμε όρια αγορεύσεις 5 λεπτά να υπάρξει χρόνος για συζήτηση. Και για μια μισή ώρα θα συζητήσουμε ε, σαν πάνελ για το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας όσον αφορά τις εκλογές και την ευρωπαϊκή η ιδιότητα του πολίτη. Αλλά επίσης θα συζητήσουμε και τα του εκλογικού νόμου του 76 που αφορούσε τις ε, ευρωεκλογές, τη εθνική δημοκρασία, την έννοια που έχει ε, στο δημοκρατικό μας σύστημα και το θέμα της αναβάθμισης της συμμετοχικής δημοκρατίας που αποτελεί το αντικείμενο της ε, γνωστής πρωτοβουλίας. Πρώτα-πρώτα έχουμε τα εκλογικά δίκαια για όλη την Ευρώπη. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ ε, περίπλοκα και υπάρχουν διάφορες επιλογές που πρέπει να γίνουν οι οποίες είναι δύσκολες, είναι πρόκληση και αφορούν τις ευρωεκλογές και πολλές φορές όμως ξεχνούμε. Ξεχνούμε το ότι σε σχέση με Ευρωπαϊκή τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι ορίζει ε, η συνθήκη και λέει ότι θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα των ευρωεκλογών. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο σύστημα ή να υπάρχουν τέλο πάντων κοινέ αρχέ για όλα τα ε, κράτη-μέλη και είπαμε ότι ακόμη δεν έχουμε πετύχει πλήρως αυτόν τον στόχο διότι οι ευρωεκλογέ διαπονται ακόμη από τα εθνικά εκλογικά δίκαια και κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική προσέγγιση. Και οπότε ε, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στην προσέγγιση το οποίο έχει σχέση με το θέμα της ιδιότητας του πολίτη και της ισότητας όπως αυτά ορίζονται από τη συνθήκη και αυτές οι διαφορές είναι κάτι το περίπλοκο και προσβάλλουν όμως την αρχή της ισότητας οπότε θα πρέπει τώρα να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το εκλογικό νόμο για την Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο οι πολίτες, να εμπλακούν περισσότερο. Θα πρέπει να υπάρξει λιγότερη αποχή. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η σημερινή εικόνα των πραγμάτων. Επίσης θα πρέπει να συμβάλλουμε στο πώς θα υπάρξει πραγματικά ε, ο Δήμος, το, το, το, το μια ευρωπαϊκή σφαίρα όπου να αναπτύσσεται ε, η εκλογική προβληματική, και έτσι επομένως θα πρέπει να έχουν περισσότερη ποιότητα στην οργάνωση των εκλογών, ε, ισότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και όλα αυτά είναι στόχοι σε σχέση με την μεταρρύθμιση για το εκλογικό μας σύστημα. Αυτό σας τονίζω και το τονίζω και πάλι θέλουμε με μια πρόταση όχι να έχουμε κάποιο είδους πλήρη ε, ομογένεια, ομοιογένεια, αλλά θέλουμε να ε, έχουμε περισσότερη ε, ισορροπία, λογική και ε, τέτοιες λύσεις να προτείνουμε όσον αφορά τις προτινόμενες διαδικασίες σε αυτόν τον εκλογικό νόμο και να συνεχίσει βέβαια να υπάρχει περιθώριο δικρατικής ευχέρειας για τα κράτη-μέλη και αυτό καλύπτει και το Συμβούλιο για διαφορετικά του. Οπότε και υπάρχει αυτό το σχέδιο εκλογικού νόμου από δύο εισηγητές, από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες και έτσι αρχίζει ε, και η συνεδρίαση με τον συνόδο με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Είναι ο Γιώ Λάινεν. Έχεις τον λόγο για μόνο πέντε λεπτά, Γιώ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίζω όλους όσοι ήρθαν σε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Δεν έχω πρόβλημα με τα πέντε λεπτά, γιατί λίγο πολύ είπατε τα ώρα. Περιλαμβάνει η πρόταση, την οποία και περάσαμε με πτυχία από την Επιτροπή ΑΦΚΟ και πλέον θα περάσει την Ελομέλεια. Δεν ήταν και εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει το πετύχαμε και θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε συγχαρητήρια στους εαυτούς μας, γιατί το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου εφαρμόστηκε με την πρόταση αυτή. Και πιστεύω ότι όλοι εδώ συμφωνούν ότι η συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έζησε μια σημαντική στιγμή και κάθε πέντε χρόνια ε, εκλέγουμε το μοναδικό πολυεθνικό κοινοβούλιο στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα που να προσωμιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε το μοναδικό κοινοβούλιο το οποίο εκλέγεται άμεσα και ελεύθερα πέρα από τα εθνικά σύνορα. Αλλά ήταν και η πρώτη φορά που συμμετείχα στην προεκλογική. Μάλλον ε, από όλε τι φορέ που συμμετείχα σε προεκλογική εκστρατεία πρέπει να πω ότι πάντα ελπίζω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά ουσιαστικά επιδεινώνεται. Στι ευρωεκλογέ, λοιπόν, έχουμε εθνική προεκλογική εκστρατεία, εθνικέ συζητήσει, εθνικού καταλόγου και υπάρχει και όλο και πιο πολύ εθνικισμό. Άρα όλα τα θέματα τα ευρωπαϊκά τα κοιτάμε από εθνική σκοπιά, ακόμα και στις ευρωεκλογέ. Ένα αυτό είναι καταδικασμένο σε αποτυχία και από την χάνει. Άρα λοιπόν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μεταρρυθμίσουμε τους όρους αυτούς για να είναι πραγματικά ευρωπαϊκές οι εκλογές. Προτείναμε λοιπόν και ξέραμε ότι ήταν πολύ φιλόδοξη η πρόταση να μπορεί το Συμβούλιο να αποφασίσει με ομοφωνία για την ε, καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής περιφέρειας. Και έτσι λοιπόν να εκλέγονται τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις χώρες το είχαμε ζητήσει αυτό ήδη πριν από 20 χρόνια. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, ότι θα υπήρχαν πολλέ αντιρρήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήταν και το καθοριστικό. Αυτό θα ήταν και το μεγάλο επίτευγμα, να γίνει μια ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία, μια προεκλογική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συμφωνούν τα ευρωπαϊκά κόμματα σε ευρωπαϊκού καταλόγου που θα ε, ψηφίζονται από όλου του πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν λοιπόν ε, πραγματικά κορυφαίο επιτεύγμα, αλλά ξέρουμε ότι είναι και πολύ φιλόδοξο. Δεν είχαμε την σχετική ευκαιρία για το 2019. Προτείναμε λοιπόν οι κορυφαίοι υποψήφοι για τα ευρωπαϊκά κόμματα να εκλέγονται τουλάχιστον 12 ε, εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών. Νομίζω ότι σημειώθηκε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός το 2014 και θα πρέπει να επαναληφθεί αυτό το 2019 και ξέρουμε ότι ακόμα και σε αυτό υπάρχει μεγάλη αντίσταση γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν πραγματικά ε, να υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση, δεν θέλουν να υπάρχουν και ευρωπαίοι κορυφαίοι υποψήφοι. Το Συμβούλιο αντιστέκεται και συζητάει την πρόταση αυτή. Τρίτο θέμα το θέμα προβολής των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ήμουν ε, το 2003 εισηγητής για τον κανονισμό, ισχύει λοιπόν 13 ε, χρόνια, αλλά δεν μπορούν να δράσουν ουσιαστικά γιατί δεν ε, υπάρχει αρκετή προβολή. Προτείνουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, ακόμα και στα ψηφοδέλτια, εκεί που γίνεται αναφορά του Εθνικού Κόμματος, να υπάρχει και παράλληλη αναφορά των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων και σιγά σιγά να τις ε, μάθει και ο πολίτης. Αυτό είναι βασικό στοιχείο θεωρώ για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση των ευρωεκλογών. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω. Η διαφάνεια και το πόσο σημαντικό είναι να προετοιμάζονται σωστά οι ευρωεκλογέ. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι από κράτος μέλος σε κράτος μέλος από 17-95 ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών ε, υπάρχει διακύμανση για τους ε, υποψηφίους. Ε, μα πώς μπορεί να κάνει κανείς προεκλογική εκστρατεία όταν μαθαίνει ότι πρόκειται να είναι υποψήφιος 17 ημέρες πριν από τις εκλογές. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτά ποιο θα κάνει. Το, η γραμματεία των κομμάτων τελευταία στιγμή και ο πολίτης τελικά δεν ξέρει καν ποιοι είναι οι υποψηφοί του γιατί δεν ε, έχει την ευκαιρία να τους γνωρίσει. Είπαμε λοιπόν ε, να ορίσουμε 12 εβδομάδες πριν τις εκλογές ως καταληκτική ημερομηνία. Τρεις μήνες δηλαδή. Αλλά Αλλά τις δύο-τρεις εβδομάδες πριν δεν έχει νόημα, δεν είναι σοβαρή η πρόταση αυτή και αυτό καταδεικνύει ότι η πολιτική ελίτ δεν μπαίνει στα σοβαρά τις ευρωεκλογές, αυτό θέλουμε να τα αλλάξουμε. Για την ισότητα, θέλουμε ισότητα μεταξύ των φίλων υπάρχει ήδη καλή εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι επαρκή αυτή η εκπροσώπηση. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό, είναι το ίμεση τη κοινωνία άλλωστε οι γυναίκε. Αλλάζοντα λοιπόν το, την εκλογική νομοθεσία, σε τελική ανάλυση αυτό θα σημαίνει ότι θα υπήρχε πίεση προς τα πολιτικά κόμματα να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ των φύλων. Κάναμε λοιπόν τη δουλειά μας, ε, το Κοινοβούλιο και η Ολομέλεια ότι είχε να προτείνει. Τώρα πλέον το μπαλάκι είναι στην πλευρά του Συμβουλίου. Ξέραμε ότι χρειάζεται ομοφωνία. Και πάντα φυσικά κάποια χώρα είναι αντίστοιχη. Και άρα στην τελική ανάλυση ε, έλαβε ο κίνδυνο να μην προκύψει τίποτα ω αποτέλεσμα. Θα ήταν μεγάλο κρίμα αυτό. Και με την κοινωνία των πολιτών και με την βοήθεια όλων σα θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, θεωρώ, να δημιουργηθεί αυτή η ορμή, αν θέλετε, προκειμένου να έχουμε ρεαλιστικές προτάσεις από επόμενες ευρωεκλογές, να βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί ντρέπομαι για το γεγονός ότι ακόμα και αν οι πολιτικοί και τα κόμματα πάντα υπερασπίζουν την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή διάσταση κτλ. κτλ αλλά όταν ε, πρόκειται να λάβουν μια συγκεκριμένη απόφαση, είναι έτοιμοι και έχουν έτοιμο το επιχείρημα του γιατί δεν γίνεται. Ας ασκήσουμε λοιπόν πίεση για να έχουμε καλύτερους όρους και συνθήκες για πραγματικά ευρωπαϊκές εκλογές το 2019. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Γιώ Λάινεν. Όχι, επτά λεπτά μίλησε. Ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Χουαρεγγί. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει στην ΑΦΚΟ που έχει βεβαίως σχέση με όλη τη συζήτηση πολιτικού περιεχομένου που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μιλήσω για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Είχα την ε, τιμή, την τύχη να είμαι εισηγητής της έκθεσης «Η Δημόκραση» που έχει ως στόχο να συνδέσει την ε, δημοκρατία με όλες τις νέες ε, τεχνολογίες επικοινωνίας που μας προσφέρονται και που μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερη τη δημοκρατία. Η βάση της ε, συζήτησης που έχουμε αφορά τη δική μας τη δημοκρατία γενικότερα. Αναφέρομαι στην Ευρώπη και όλα τα κράτη της μέλη. Και βλέπουμε ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα που μας επιτρέπει να πούμε ότι έχουμε δημοκρατική κρίση. Μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο με πολλούς τρόπους. Εμείς είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αναφορά στο θεώρημα του Ρόντρικ. Δηλαδή όσο περισσότερη παγκοσμιοποίηση τόσο λιγότερη δημοκρατία έχουμε. Δεδομένου ότι βασίζεται η δημοκρατία πολύ περισσότερο στο κράτος έθνος και στην παγκοσμιοποίηση έχετε δυσκολίες ε, αυτό το πράγμα να το δείτε να εφαρμόσετε και ιδιαίτερος το βλέπουμε στην Ευρώπη. Γιατί μιλούμε για δημοκρατική κρίση. Διότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη δυσκολία να εξηγήσουμε την πολυπλοκότητα της διακυβέρνησης και στους πολίτες να δώσουμε να καταλάβουν πόσο πολύπλοκε είναι οι αποφάσει που πρέπει να λαμβάνουμε. Μιλούμε για κρίση διότι υπάρχει δυσπιστία στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα ή αδιαφθορά ή για άλλα θέματα. Μιλούμε για κρίση διότι υπάρχει απομάκρυνση των ε, δημοσίων εκπροσώπων από τους πολίτες. Μιλούμε για κρίση διότι τα πολιτικά κόμματα ή θέλουν ε, αποκλειστικά να μονοπολίσουν ή να πάρουν τον εαυτό τους, αν θέλετε, την σχέση με τα θεσμικά όργανα. Μιλούμε για κρίση του θεσμικού προτύπου που υπερίσχυσε το δεύτερο ήμις του 20ου αιώνα που ήθελε να βρίσκονται σε σχέση οι πολίτες με το κράτος τους. Να έχουν σχέση διότι περιμένουν κάτι από το κράτος. Και έτσι εκφράζει θυμό ο κόσμος ε, θυμό, δεδομένου ότι έχουμε κρίση και οι συνέπειες είναι σοβαρές, διότι δεν λειτουργούν καλά δημοσιοπηρεσίες, διότι η οικονομική πολιτική σε σχέση με τις αγορές έχει τους περιορισμού της, θα ήταν ατελείωτος ο κατάλογος που θα μπορούσα να σας απαριθμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως λοιπόν επιβεβαιώνεται και πάλι ότι έχουμε ασθενή δημοκρατία. Το δεύτερο μέρος του ερωτήματος είναι η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει. Προφανώς ε, δεν έχουμε την πρόθεση με την ε, ε, έκθεση αυτή να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες λέγοντας ότι πρόκειται πράγματι για την πανάκια που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έχουμε ουσιαστικά προβλήματα προβλήματα δομικά. Αλλά μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια πολιτική, ένα πολιτικό ε, συλλογισμό και μια μελέτη για να δούμε αν με τους μηχανισμούς και τα νέα όπλα που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες μπορούμε να βελτιώσουμε τη δημοκρατία. Τελειώνοντας κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι συντάξαμε και ασχολούμε με αυτή την έκθεση όχι προσπαθώντα να καινοτομήσουμε στα πάντα, διότι πρόκειται για ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε όλοι, καθώ και άλλα θεσμικά όργανα που από το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ και 10 χρόνια. Σκέφτομαι τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι έχουν κάνει διάφορε χώρε σε σχέση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την ε, ε, συμμετοχή των πολιτών, με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με τους μηχανισμούς διαφάνειας για την διακυβέρνηση. Εγώ απλώς ταπεινά θα ήθελα να πω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, να προσφέρουμε. Αναγνωρίζοντας τι έχει γίνει και προσπαθώντας με νέες προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται για θεωρητική συζήτηση, διότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και συνεισφορές εκ μέρους και ακαδημαϊκών, πώς θα μπορέσουμε με συγκεκριμένους τρόπους και φόρμουλες να συνεισφέρουμε ώστε το σύστημα το ευρωπαϊκό και τα κράτη-μέλη μας να βελτιώσουν και το θέμα της διασύνδεσης των πολιτών με τον ε, πολιτικό κόσμο. Και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται, ξέροντας βεβαίως ότι και ε, πολλά από τα ευρήματα που έχουν γίνει μας επιτρέπουν να δούμε τι από αυτά τα οποία λέγονται είναι μύθος γιατί κάποιοι πιστεύουν ε, ότι πραγματικά οι νέες τεχνολογίες είναι η θαυματουργή λύση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, παραδείγματα που μας αποδεικνύουν ότι πολλές φορές η διαφάνεια χρησιμοποιείται περισσότερο από ομάδες συμφερόντων παρά από τους πολίτες. Και τελειώνοντας και πάλι επαναλαμβάνω κυρία Πρόεδρε, το σχέδιό μας είναι να περιχαρακώσουμε αυτά τα, αυτούς αυτά τα πλαίσια, ώστε να μπορέσουμε μέσω διαφόρων πράξεων να βελτιώσουμε την δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γιώργη Σέπφλιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω. Για τα θέματα αυτά που μου με του Ευρωπαίου πολίτη σε σχέση και με ε, την πρωτοβουλία των πολιτών για μένα η ιδιότητα του πολίτη και η ηθαγένεια σημαίνει το να έχει ρυθμιστεί η σχέση μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κακή και πρόβλημα συστήματα μας οδηγούν δυστυχώ στη δεύτερη διαπίστωση και το ιδιώδες είναι όταν μπορεί να συμβάλλει <clears throat> σαν άσκηση εξουσίας ο πολίτης και ανταποκρίνεται σε αυτή τη συμβολή εξουσία. Άρα επομένω θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, πρώτα για μια δυναμική διαδικασία γιατί και οι δύο πλευρές μπορούν κάτι να μεταβάλουν στον τρόπο της ανταπόκρισης του ενός προς τον άλλο. Τώρα, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και στον αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών, πρόκειται για ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εμπλοκή των πολιτών στις υποθέσεις Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σε σχέση και με τις εξουσίες ομότητες αυτές. Ας μην επιστρέψουμε στις λεπτομέρειες, όλα αυτά κατοχυρώνονται στην συνθήκη στο άρθρο 11 παράγραφος 4 και είπαμε ότι με ένα εκατομμύριο υπογραφέ για οποιοδήποτε θέμα ε, είναι δυνατόν να θεσπιστεί κάποια νομοθεσία και κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι αποδυναμώνεται το μονοπόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη θέσπιση κάποιου νόμου και υπάρχει εδώ μια δυνατότητα, μια πολύ βασικό εργαλείο. Παρόλα αυτά ε, τέσσερα χρόνια ε, που τρέχει αυτή η πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θέλετε μεγάλο ή μικρό διάστημα. Βλέπουμε ότι έχουμε εδώ πέρα ε, διάφορες τις πρωτοβουλίες που έχουν ε, αναπτυχθεί, κάποιες έχουν γίνει αποδεκτές, κάποιες είναι ακόμα στη φάση της συλλογής υπογραφών, από ό,τι γνωρίζω δεν έχουμε κάτι τώρα πιο πρόσφατα, αλλά ούτε μία πρωτοβουλία δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο, δηλαδή σε νομοθέτημα. Άρα νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι ένα πετυχημένο εργαλείο η πρωτοβουλία των πολιτών. Και τι λένε οι επισόδους, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Απέτυχε η πρωτοβουλία. Εγώ όμως δεν είμαι πιο δεν λέω ότι απέτυχε, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και καμιά τρομερή επιτυχία, γιατί ακόμα επιδέχεται μεγάλες βελτιώσεις και από την Επιτροπή. Εδώ στο Κοινοβούλιο παρακολουθούμε τι γίνεται στην ε, ΑΦΕΤ συγγνώμη, στην ΑΦΚΟ, την Δημοτική Επιτροπή και είπαμε ότι με βραδύ τρόπο έχει αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το πω διπλωματικά και έχουμε την αρχική αντίδραση που δεν ήταν και τόσο ε, αποτελεσματική και από τον κόσμο ακούγεται ότι χάνετε το χρόνο σας λένε ακόμα μπορούν να βελτιώσετε κάτι, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει η Κομισιόν να έχει άλλη αντίδραση. Αυτό το λέει ο κόσμος, αυτοί που έχουν εμπλακεί. Δεν έχω ακόμα στοιχεία για το πόσες προγραφές έχουν πέσει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για, πάντως για κάποια εκατομμύρια. Πάρα πολλοί από αυτού λένε ότι τίποτα δεν θα βγει, χάνουμε το χρόνο μας. Γιατί να το κάνω αυτό για να μην ήμουν ευρωσκεπτική στις ε, δεν είναι και τόσο παράλογο έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτό το οποίο λένε και εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια να αποδώσει αυτό το εργαλείο, πρέπει να κάνουμε και άλλα και θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτή εξουσία ε, σε όλα αυτά που ακούγονται από τον κόσμο, σε αντιδράσει του κόσμου. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, βέβαια, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Τη υπηρεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ο Πολ Νέμιτσα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ γιατί φυσικά όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ε, δημοκρατία στην Ευρώπη και πρόκειται για μια ε, επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτε άμεσε εκλογέ του 1979, στην το θέμα της ε, των κορυφαίων υποψηφίων ήταν ε, θέμα πολιτικής, ε, πολιτικού επιτεύγματος και χρειάστηκε ουσιαστικά δύο δεκαετίες για να περάσει αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο το οποίο υποστήριξε και παρουσίασε ο Γιώ Λάινεν, το υποστηρίζουμε. Είναι μια προσπάθεια κωδικοποίηση του κορυφαίων αυτών υποψηφίων προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα η δημοκρατία. Πρόκειται για μία μάχη για το καλύτερο λοιπόν, μία ε, ιστορία επιτυχίας, αλλά έχουμε και πολλά να κάνουμε. Θα ήθελα να σα δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία και κάποια γενικότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αυτή βάσει του πρόσφατη μελέτη και έρευνα. Υπενθυμίζουμε την προσέλευση στι τελευταίε εκλογέ με τους κορυφαίους αυτούς υποψηφίου. Πού είναι λοιπόν τα οι αν θα μπορούσατε να τι προβάλλετε παρακαλώ στην οθόνη, μάλιστα την δεύτερη οθόνη περάστε. Την δεύτερη διαφάνεια. Να σα υπενθυμίσω λοιπόν ότι με την εισαγωγή των κορυφαίων υποψηφίων η σαφέστατη καθοδική τάση στην προσέλευση έλαβε τέλος και μόνο 0,39% ήταν η καθοδική τάση αυτή. με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στη συμμετοχή στην προσέλευση. Πολύ χαμηλή προσέλευση, ιδιαίτερα στις νέες χώρες μέλη, στην Ανατολική Ευρώπη. οι λόγοι τώρα γι' αυτό. Ενδεχομένω ε, το εθνικό κλίμα σε ό,τι αφορά την δημοκρατία να καθορίζει και την ε, συμμετοχή στι ευρωεκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει εκθέσει και μελέτε για τη συμμετοχή των πολιτών και στι εθνικέ εκλογέ. και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή την τάση και εκεί. Άρα η χαμηλή προσέλευση στις ευρωεκλογέ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη. το θέμα της χαμηλής συμμετοχής στις εκλογές διαπιστώνεται σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στο τοπικό δημοτικό επίπεδο. Άρα το κλασικό επιχείρημα ότι οι πολίτες δεν θέλουν την Ευρώπη και δεν καταλαβαίνουν την ε, Ευρώπη δεν ισχύει, δεν στέκει, γιατί και στο τοπικό επίπεδο έχουμε πολύ χαμηλή προσέλευση. Τώρα, να σας δείξω αυτό που αποκαλώ τα μικρά και τα μεγάλα θέματα της δημοκρατίας. Τα μικρά θέματα της δημοκρατίας. 40 εκατομμύρια ε, κράτη, ε, Ευρωπαίοι πολίτες που μένουν ε, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν, ξέρουν τι μπορούν να ψηφίσουν και λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και έτσι θα περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο και εγώ θα σας λέω πάντα που βρισκόμαστε. Στη διαφάνεια λοιπόν αυτή που βλέπετε τώρα κοιτάμε τα μικρά ζητήματα της δημοκρατίας. Ξέρει ο κόσμος, για παράδειγμα, ότι οι πολίτες που διαμένουν σε άλλη χώρα έχουν δικαίωμα ψήφου. 40 εκατομμύρια. Οι απο... απαντήσεις είναι σχετικά ακριβείς. 67% το γνωρίζει ότι μπορεί να ψηφίσει και από άλλη χώρα. Στην επόμενη διαφάνεια περνάμε πάλι σε μεγάλο ζήτημα της δημοκρατίας πώς μπορούμε να βγάλουμε τα 400 εκατομμύρια ψηφοφόρους στις κάλπες. Δεν βλέπουμε κάτι ε, που να μας προκαλεί έκπληξη. Φυσικά, ο κόσμος θέλει να ξέρει κατά πόσο τον αφορούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, κατά 84% προγράμματα και στόχοι των υποψηφίων και ε, στοχοθέτηση των κορυφαίων υποψηφίων, 77%. Αυτό είναι σημαντικό. Καταδεικνύει ότι είναι σημαντικό το θέμα του κορυφαίου υποψηφίου και επίσης ε, αναφέρεται ότι στην 72% θέλει να υπάρχει κάποια σχέση με το προεκλογικό υλικό. Πάμε πάλι στην επόμενη διαφάνεια για τα μικρά θέματα να κοιτάξουμε. Είναι πολύ ρυθμική αυτή η παρουσίαση. Πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. 21% των πολιτών έχουν περάσει δυσκολίες ε, όταν ήθελαν να ψηφίσουν ε, από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πάλι μιλάμε για τα 40 εκατομμύρια. 51% λοιπόν των 40 εκατομμυρίων θεώρησε ότι είχε προβλήματα για να ψηφίσει από άλλη χώρα. Αυτό για την για το μικρό θέμα της ε, συμμετοχής στις ευρωεκλογέ από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα, μιας και συζητάμε δικαιώματα του πολίτη, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και ξανά στην επόμενη διαφάνεια πάμε σε ένα μεγάλο θέμα της δημοκρατίας. Η άποψη των πολιτών για το τι θα μπορούσε να διευκολύνει την ψηφοφορία σε ευρωπαϊκέ. Α, συγγνώμη, αυτό είναι μικρό ζήτημα. 40 εκατομμύρια, φορά. Άρα, τι λέμε ο 80% πιστεύει ότι καλά θα ήταν να υπήρχαν μεμονωμένε επιστολέ που την εξηγούν. Και μια αυτόματη καταχώρηση. Στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε πάλι σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ζήτημα. Πιο πολύ πρόσβαση στι ειδήσει και στι πολιτικέ ε, συζητήσει ε, πέρα από τα σύνορα. Να σα πω ότι αυτό που είδαμε με του κορυφαίου υποψηφίου στην προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία ήταν το εξή. Καταρχά, μεγάλη δημοσιότητα. Απίστευτη δημοσιότητα έλαβαν αυτοί οι υποψήφοι όταν ταξίδεψαν και μεγάλη καθοριοποίηση και στα κοινωνικά μίλια. Όταν όμως έγιναν οι, τα debate, η μετάδοση των ε, debate αυτών ήταν σε κάποιες περιπτώσεις ε, με γεωγραφικό αποκλεισμό πρόβλημα αυτό και θα προσπαθήσουμε αυτό να το επιλύσουμε στους κανόνες για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Προκειμένου στο μέλλον όταν γίνονται πολιτικά debate που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές πληροφορίες να μην υπάρχει γεωγραφικός αποκλεισμός. Σημαντικό αυτό. Όχι μόνο για τις ευρωεκλογέ, προκειμένου να παρακολουθεί ο κόσμος τις συζητήσεις μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων, αν γίνει στην Ιταλία δηλαδή η συζήτηση, να μπορεί να τη δει όλο ο κόσμο. Αλλά αυτό είναι σημαντικό για τη δημοκρατία και στο ιστορικό των κρατών μελών. Πάρα πολύ ουσιώδη αυτή η μετατροπή. Θα πρέπει να υπάρχει μετάδοση πέρα από τα όρια των συνόρων. Και στην, σε ό,τι αφορά την ε, τα μέσα ενημέρωση. 53% λοιπόν δήλωσαν ότι ήταν εν μέρη ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες που έλαβαν. Αλλά σχολιάστηκε το θέμα του γεωποκλεισμού. 83% θα ενδιαφέρονταν για να έχουν πρόσβαση σε πιο πολλά προγράμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 90% πιστεύουν ότι αυτή η καλύτερη πρόσβαση θα τους επιτρέπει να σχηματίσουν καλύτερη πολιτική άποψη. Τέλος, ε, τελευταία διαφάνεια, να σας υπενθυμίσω, όχι κάτι καινούριο, μία υπενθύμηση ότι σε πολλά από τα κράτη-μέλη, το διαδίκτυο και τα κοινωνικά media, Google, Facebook και Twitter, έχουν καταστεί υπαρισμόν ένα πηγή για πολιτικές πληροφορίες. Και αυτό μας απάντησαν και οι ερωτηθέντες, ότι πλέον βασική πηγή είναι το διαδίκτυο, πάνω από 70% και τα κοινωνικά ε, 50% παραπάνω Άρα, από κοινού είναι πολύ πιο σημαντικές πηγές σε σχέση με τις εφημερίδες και τη τηλεόραση. Άρα, όταν σκεφτόμαστε πολιτικές ειδήσει και πολιτική ενημέρωση, πρέπει να σκεφτόμαστε ίντερνετ και κοινωνικά μέσα. Και τελευταίο σημείο, το τι αφορά την κινητοποίηση, σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση της ε, κοινή γνώμη, δεν φτάνει να το κάνουμε αυτό την ημέρα των εκλογών. Ας δείξουμε διαρκώς με ποιο τρόπο μπορούν οι Βρυξέλλες να οδηγήσουν σε αλλαγή. Και να σας πω ένα παράδειγμα, τέσσερα παραδείγματα μάλλον για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πρόσφατη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων. Το αποτέλεσμα, τι θα ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχαν 20 ακτιβιστή, όπως ο Μάξ Φέντς από τη Βιέννη ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για να αντιμετωπίσει το λόμπι των μεγάλων εταιριών. Νομίζω ότι τέτοιου είδου επιτυχίε και τον εξηγήσει και ποιο ήταν ε, ο κόσμο, ο άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την επιτυχία αυτή. Αυτά πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εμβληματικά από όταν αναφέρει κανεί ε, την τάδε ή νομοθεσία και το καλό είναι ότι αυτό αποτυπώνεται και στα δικαστήρια και τα δικαστήρια ανταποκρίνονται στι ανάγκε του πολίτε. Ο Μαξ Σρέμ έλαβε μια σημαντική δικαστική απόφαση σε ό,τι αφορά το ασφαλή λιμένα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την κράτηση των προσωπικών δεδομένων και βλέπουμε λοιπόν ότι τα δικαστήρια ανταποκρίθηκαν στι ανάγκε τη κοινωνία των πολιτών και το κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο δεσμεύτηκε δεσμεύτηκαν κάποιοι Και αυτό σημειώνει τη διαφορά. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να προβάλλουμε καλύτερα αυτές τις επιτυχείς ιστορίες προς τους πολίτες. Και αυτό να γίνεται διαρκώς, όχι μόνο την ημέρα των εκλογών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διευθύντη Νέμιτς, και να σας πούμε ευκαιρία ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Κομισιόν στην διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ριντάφ, πρώην συνάδελφός μας και έναν ένα από του πιο Ευρωπαίου Ευρωπαίου. Έχετε το λόγο, Άντριο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη ευχαρίστηση είμαι εδώ και θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές που ασχολούνται με το θέμα της αναθεώρησης του εκλογικού νόμου Πρέπει να πω ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι φαίνεται και πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι πιστεύουμε. Και βεβαίως γνωρίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα ρε, του Κοινοβουλίου. For the commission to, uh, to be asked to... Όπως γνωρίζουμε, έχει ζητηθεί από την Επιτροπή και φέτος να κάνει μία πρόταση και βεβαίως είναι με ευχαρίστηση για το Συμβούλιο να περιμένω του υποβάλλουν την πρόταση να χρειαστεί να το κάνει μόνο του. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για πολύ μεγάλη δημοκρατική κρίση στην Ήπειρό μας. Πρόκειται για αποτυχία των εθνικών πολιτικών κομμάτων να συνεχίσουν να εξηγούν ή να δικαιολογούν το γιατί πρέπει να υπάρχει ενοποίηση. Κάποιοι έχουν εγκαταλείψει τέτοιου σχέδια, κάποιοι αγνοούν περί την πρόκειται, κάποιοι άλλοι ζηλεύουν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως κάποια εθνικά πολιτικά κόμματα έχουν μια εντελώς αρνητική προσέγγιση όσον αφορά θέματα σημαντικά όπως αυτό της αντιμετώπισης των προσφύγων. Ο κύριος στόχος τον οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε είναι να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε ή κατά κάποιο τρόπο να δώσουμε μία πολιτική διάσταση σε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κόμμα τα, για τέτοιου είδου θέματα δημοκρατίας συμπληρώνοντας τις δράσεις των εθνικών πολιτικών κομμάτων. Ξέρουμε βεβαίως ότι κάποιοι αγωνίζονται για να έχουν εκείνα και την πολιτική εξουσία και να έχουν περισσότερη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποφασίζουν για τις πολιτικές. τα αποτελέσματα της ε, μίζης της δημασίας των ε, εθνικών κομμάτων το βλέπουμε όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα των ε, εκλογών. Υπάρχει πολύ λίγη ανταπόκριση εκ μέρους των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά το θέμα της αναθεώρησης της εκλογικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να πω ότι έχουν υπάρξει διάφορες αντιρρήσεις εκ μέρου των Εθνικών Κοινοβουλίων στι προτάσει που κάνουμε εμεί για την μεταρρύθμιση τη εκλογική διαδικασία. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να, ό,τι γίνεται να το λαμβάνουμε υπόψη και να τους εξηγήσουμε πότε εφαρμόζεται η επικουρικότητα και με ποιο τρόπο κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και να απαντήσουμε στις επικρίσεις του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο παρελθόν που γνωρίζω καλά εγώ, αλλά και σήμερα δεν μπορεί πολλές φορές να εξηγήσει ή να αιτιολογήσει τις προτάσεις που υποβάλλει. Παρά το γεγονό ότι το σχέδιο απόφασης προσπαθεί να διασυνδέσει έτσι όπως περιγράφεται αυτό που λέμε κοινή εκλογική περιφέρεια με τον Spitzen Candidat δεν γίνονται αξιόλογες και επαρκείς εξηγήσει ώστε να υπάρξει σε επίπεδο διαλόγου μεταξύ των τριών οργάνων διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνίες γενικά. Βεβαίως, σωστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να βελτιώσει ό,τι αφορά αυτή την διαδικασία του speech and candidate. Αλλά υπάρχει και το θέμα της κατανομής των ευρών στον πρωτογενές κοινωτικό δίκαιο. Ξέρουμε ότι έχουν ε, αλλάξει κάποια πράγματα που έχουν κάνει το κοινοβούλιο να χάσει ίσως σε κάποια θεσμική φύσεως θέματα την νομιμοποίησή του. Κάποια μέλη λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσπαθούν να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο της όλης διαδικασίας εκλογής του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό. που έχει σχέση με απόφαση που ελήφθη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι όπως εξηγείται στην έκθεση Verhofstadt. που αναφέρεται στις αλλαγές τις οποίες θα επιθυμούσε να δει να γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επόμενη συνέλευση θα μπορούσε να προβλέψει ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία πρώτα απ' όλα όσον αφορά την εκλογική διαδικασία καθώς και συμφωνία σε άλλα θέματα όπως φερειπίν το θέμα της ε, αλλαγής του τρόπου κατανομής των θέσεων. Και λήψη. μια ε, πλήρους συνθήκης. Ελπίζω δε το Κοινοβούλιο πλέον να επικεντρωθεί στην προετοιμασία για, μια τέτοια, για ένα τέτοιο εγχείρημα. Να προετοιμαστεί λοιπόν το Κοινοβούλιο για να επηρεάσει τις μεθόδους εργασίας, της ε, συνέλευσης, της συνθήκης και να προετοιμάσει και το έδαφος, να προλειάνει το έδαφος για τις ε, διαπραγματεύσεις επί της ουσίας που θα λάβουν χώρα. Σε ό,τι αφορά το timing δε, όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε φαντάζομαι δυστυχώ ότι αυτό δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν τις ευρωεκλογές σε Τρία χρόνια. Είναι όμως απαραίτητο η άσκηση αυτή, η απόπειρα να ενισχυθεί και να ευανθυθεί. Η άσκηση της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο θα παίξει σημαντικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες. στις ε, προεκλογικές εκστρατείες των πολιτικών ομάδων, αλλά και του Κοινοβουλίου γενικότερα. Και θα λειτουργήσουν ως μία άδεια για μία πιο ενημερωμένη και τεκμηριωμένη εκστρατεία. πιο πολύ από ό,τι έχει πετύχει έω τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άντριου. Θα ήθελα τώρα να έχει έρθει ο Ιβ Μπεθοντσίνη. Α, έχει φτάσει. Ε, πρέπει να σας ενημερώσω και εσάς. Πέντε λεπτά παρακαλώ έχετε στη διαθέσή σας. Είστε διευθυντής του Ινστιτούτου Ζακ Ντολό. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με μπλοκάρανε στην είσοδο. Συγγνώμη λοιπόν που καθυστέρησα. Ας έρθω στο θέμα μου. Σας έχω αφήσει κάποια έγγραφα στην είσοδο της αίθουσα για να τα συμβουλευτείτε. Κάποιες πολύ γρήγορες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όταν ασχολούμαστε με την ε, ηθαγένεια και την συμμετοχή τους και τι σημαίνει αυτό, να κάνουμε κάτι το ποιοτικό. Ας σκεφτούμε το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ποιο είναι. Όπως στην Ελβετία και στη ΣΥΠΑ. Γύρω στο 40 με 50% γιατί και το κράτος και ο Δήμος δεν είναι έννοιες που έχουν μεγάλη σημασία. Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε με μια πιο ποιοτική προσέγγιση να κάνουμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κάνουν κάποιες επιλογές όταν ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και είναι χρήσιμο και για αυτούς να βλέπουν και τα πρόσωπα των ατόμων τα οποία θέλουν να ψηφίσουν. Τώρα, το θέμα αυτού των Spitzenkandidaten είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να μελετήσουμε. Είδαμε τι έγινε το 2014 και θέλουμε να προχωρήσουμε και περισσότερο. Διότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημα και να δώσουμε στα πολιτικά κόμματα περισσότερα μέσα δεδομένου ότι είναι ο αδύναμος κρίκος μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών δεσμών. Περισσότερα μέσα, περισσότερα κονδύλια, τρίτη μου παρατήρηση. Και όχι μόνο λίγα χρήματα στους πολιτικούς. Ξέρουμε ότι οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διαφορετικά από άλλα πολιτικές ομάδες. Είναι, έχουν ενηλικιωθεί πλέον, δεν τους δίνουμε όπως στα παιδιά χαρτζηλίκη. Πρέπει να τους δώσουμε περισσότερα κονδύλια, να τους διαθέτουμε. Όχι να το πάρουμε από κάποιον άλλο για να το δώσουμε, αλλά να τους δώσουμε ε, περισσότερα χρήματα διότι κοστίζει, είναι δαπανηρή η δημοκρατία. Uh, European citizens or at least European citizens. Αν θέλουμε λοιπόν να επηρεάσουμε θετικά τους Ευρωπαίους πολίτες για να κάνουν την επιλογή τους και να ψηφίσουν ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει να τους δώσουμε περισσότερα κονδύλια και να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και να επιτρέψουμε και σε άλλους φορείς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας όπως ιδρύματα ή άλλους φορείς να είναι πιο ενεργοί, πιο δυναμικοί να συμμετέχουν περισσότερο. Να καταρτίζουν και τους ακτιβιστές που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εκλογές. Και δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν θα εξαρτηθούν από τι εναλλακτικέ λύσεις που προσφέρουν για τη διάρκεια της επόμενης εκλογικής εκστρατείας. Πρέπει να πω ότι το 2004 δεν ήταν η, ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες βεβαίως, που το καθένα μπορεί να οργανωθεί όπως θέλει. Θα πρέπει για να προχωρήσουν περισσότερο τα κόμματα, να τα βοηθήσουμε, να έχουν μεγαλύτερες επιλογές και εναλλακτικέ λύσεις και να κάνουν και κάποιες συναντήσεις, συνεδριάσεις για να ορίζουν τους υποψηφίους τους και να κάνουμε και primary elections όπως έχουν και οι ΙΠΑ. Τέλο πάντων το αναφέρω για να πω ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά κονδύλια θέλουμε να προωθήσουμε και τέτοιες εναλλακτικέ λύσεις. Συμπερασματικά υποστηρίζουμε αυτά που είπε ο κύριος Νταφ. Δηλαδή, αν υπήρχε περισσότερος πανευρωπαϊσμός στις λίστες των υποψηφίων, θα ήταν ίσως τα πράγματα καλύτερα. Και αντί να δημιουργήσουμε ίσως πανευρωπαϊκές λίστες, δώσουμε οικονομικά κίνητρα ώστε ένας από τους τέσσερις υποψήφιους να μην είναι ε, υπήκος αυτής της χώρας, ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση περί ευρωπαϊκών εκλογών. Αυτά μπόρεσα να σας πω σε 5,5 λεπτά. Σας ευχαριστώ και τώρα ξαναπερνάμε στην ε, Κομισιόν Γενική Διευθύντρια, ε, η κυρία Σα σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα επανέλθω στα θέματα τα οποία σχολιάσατε ήδη και χαίρομαι και είμαι ευγνώμων προ ε, του συναδέλφου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέσατε το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι το πιο πρόσφατο ενδεχομένω δικαίωμα των πολιτών, το οποίο εισήχθη με την συνθήκη τη Λισαβόνα και εφαρμόζεται από το 2012 και μετά. Βρίσκεται λοιπόν σε μια πρώτη ε, φάση διαμόρφωσης θα προσπαθήσω να σας δώσω στα πέντε λεπτά που έχω πιο, όσο πιο πολλά α, γεγονότα και στοιχεία έχουμε για το πού δουλεύει καλά και πού δεν δουλεύει καλά η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία αυτή και πώς θέλουμε να βελτιώσουμε την διαδικασία, τι κάνουμε ήδη για να βελτιώσουμε την διαδικασία και τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον προκειμένου όλοι οι πολίτες να μπορούν να ωφεληθούν από τον εαυτό δικαίωμα, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά και να καταστεί ένα ουσιαστικό εργαλείο Συμμετοχή δημοκρατική των πολιτών. Θα ήθελα επίση να αποτελέσω στα πέντε λεπτά μου και ένα αντιστάθμισμα προς τον κύριο Σόπλιν. Γενικά ε, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την ε, ερμηνεία μας. Πέντε χρονών λοιπόν είναι αυτή η πρωτοβουλία, δεν είναι και πολύ μεγάλη. Ε, τι πάει καλά, να μην ξεχνάμε τα θετικά στοιχεία Ακούσαμε ότι έχουμε παραπάνω από 35 πρωτοβουλίε που έχουν καταχωριστεί στην Κομισιόν. Δεν έχουμε επακριβή στοιχεία σε ό,τι αφορά τι επιστολέ υποστήριξη από πλευρά των πολιτών, αλλά σίγουρα ξεπερνούν τι 6 εκατομμύρια. Τρει ήταν οι επιτυχίε τέτοιε πρωτοβουλίε που έφτιασαν το το, το ορισμένο όριο και έχουμε πέντε πρωτοβουλίε οι οποίε είναι ακόμα στη φάση συλλογή υποστήριξης για να πετύχουν ακριβώς τον στόχο και το κατόφλι, τον όριο των, του ενός εκατομμυρίου. Είναι κάτι χωρίς προηγούμενο, πρόκειται για κάτι εντελώ καινούριο και αποτελεί επιτυχία το γεγονός και μόνο ότι καταφέραμε να εφαρμόσουμε ε, τον κανονισμό. Αυτό ασφαλώς ε, δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχαζόμαστε και να μην εντοπίζουμε τα ελαττώματα, τα προβλήματα. Άρα, ελαττώματα, προβλήματα, προκλήσεις είναι πολλά. Υπάρχει μια μεγάλη διάσταση IT στη σχετική, στο σχετικό κανονισμό που προκαλεί πολλές δυσκολίες και περιπλοκότητες ό,τι αφορά τη χρήση του εργαλείου. Το ε, εργαλείο online δύσκολο στην πιστοποίηση του χρονοβόρο και αποτρέπει πάρα πολλούς πολίτες από τη χρήση του εργαλείου. Υπάρχει και το θέμα της νομικής ευθύνης. Οι επιτροπές πολιτών που οργανώνουν τις πρωτοβουλίες δεν έχουν νομική υπόσταση. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και πολλές προκλήσεις έχουν να κάνουν με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται ο κανονισμός. Να μην πεις άλλο σε λεπτομέρειε σας δίνω έτσι επιγραμματικά τον κατάλογο των βασικότερων προκλήσεων. Υπάρχει και μια μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές και τα δεδομένα. Αυτό αποτρέπει πάρα πολλούς πολίτες από την αποτελεσματική χρήση του δικαιώματο αυτού για την υποστήριξη μια τέτοια πρωτοβουλία. Και αυτό συνδέεται με το γεγονό ότι υπάρχουν διάφορε και αποκλίνουσε προδιαγραφέ για τα δεδομένα. Η αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ένα πολύ απλό σύστημα, αλλά στην πορεία των διαπραγματεύσεων κάθε κράτο μέλο του δεν λαμβάνει τα δικά του και τελικά καταλήξαμε με ένα πολύ δύσκολο και βαρύ σύστημα. Έγινε μια κοινή διακήρυξη όταν ε, εγκρίθηκε ο κανονισμό και τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να απλοποιήσουν τη διαδικασία, αλλά δεν έχουν προχωρήσει και πολύ. Αυτέ λοιπόν οι πολύ σύνθετε προδιαγραφέ για τα δεδομένα ε, αποκλείουν ένα τρομακτικό ρυθμό πολιτών από την υπογραφή τέτοιων πρωτοβουλειών. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία γιατί εξαρτώμαστε από τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Εκατοντάδες χιλιάδες όμως ε, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, που ζουν ε, στην ε, Λοδαπή, μέσα στην Ένωση, για να μην συζητήσουμε με αυτούς που μένουν εκτός Ένωσης, για παράδειγμα, Ισλανδοί που ζουν σε άλλα κράτη-μέλη. Τι κάνουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και γι' αυτό χαίρομαι που στην ακρόαση αυτή θέτουμε για το θέμα της πρωτοβουλία και αυτό είναι στα χέρια όλων των θεσμικών οργάνων να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση και την ενημέρωση για το πώς λειτουργεί το εργαλείο. Για τις προδιαγραφέ δεδομένων σας μίλησα. Ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη να απλοποιήσουν τις προδιαγραφέ αυτές για να είναι λιγότερο περίπλοκο το σύστημα και να ωφελούνται όλοι οι πολίτες από αυτό. Επίσης, στην παρούσα φάση εξετάζουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε καλύτερα την ηλεκτρονική υπογραφή. Γιατί είχαμε έκτοτε πάρα πολλέ ηλεκτρονικέ εξελίξει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά προφανώ ω τεχνολογικέ δυνατότητε. Το κάνουμε αυτό. Εξετάζουμε το θέμα αυτό εκ του συνεγγύη. Προσπαθούμε επίση να απλοποιήσουμε τι τεχνικέ προδιαγραφέ για το σύστημα επιγραμμική συλλογή υπογραφών. Όλα αυτά ένα-ένα νομίζω ότι αν τα βάλουμε όλα μαζί θα απλοποιήσουν κατά πολύ την όλη διαδικασία. Άρα, ενημέρωση, απλοποίηση και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες που θέλουν να μπορούν να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίε. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω κλείνοντα ότι το θετικό σημείο είναι ότι συγκλίνουμε με όλα τα δεσμικά όργανα, με όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των προκλήσεων και των ε, σημείων που θα πρέπει να βελτιωθούν. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν σχεδόν διαφωνίε μεταξύ Κομισιών, Συμβουλίου, ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εθνικών Αρχών για τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Υπάρχουν κάποιε διαφορέ απόψεων για το κατά πόσον χρειάζεται γρήγορη αναθεώρηση τη οδηγία ή όχι. Στην απάντηση τη Κομισιόν ε, που στέλαμε στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο, εξηγήσαμε ότι τώρα θα επικεντρωθούμε στη βελτίωση των συντημάτων που δεν προϋποθέτουν άμεση αναθεώρηση, αλλά φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πίεση και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση σύντομα. Θα περιμένουμε και την γνωμοδότηση από την Επιτροπή Οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων και επίσης το Συμβούλιο έχει ξαναξεκινήσει να συζητάει το θέμα. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν και με χαρά να σας πω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δημιούργησαν μια γραμμή στον προπολογισμό για την πρωτοβουλία των πολιτών. Δεν υπήρχε πέρσι, σας ευχαριστώ. Δυστυχώς βέβαια δεν βάλαν χρήματα στη γραμμή αυτή. Είναι μόνο μια τέτοια καταχώρηση. Αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά. Ελπίζουμε το χρόνο να έχουμε και κοντέλια. Είναι κοινή λοιπόν η προσπάθεια, κοινό και ο στόχο και νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πρωτοβουλία των πολιτών ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό εργαλείο που μπορούν να, να χρησιμοποιούν οι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων. Έχουμε μαζί μας την Ίντα Μπίρκβαλ Σόρενσεν. Ευχαριστώ. Παρουσία, εκπροσωπώντας ε, τους ε, νέους στην Ευρώπη, στην πλαίσια του Φόρουμ, εξ ονόματο πολλών εκατοντάδων νέων. αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να έχουμε μια γενιά περιστοποιημένων και χωρίς ενθουσιασμό και αυτοπάτες νέους. Η δημοκρατία δεν χτίζεται εύκολα. Πρόκειται για μια μακρόπνοη προσπάθεια για ένα δρόμο δύσκολο. 72% των νέων έχουν δικαίωμα, ε, του, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγην δεν ψηφίζουν. Πολύ λίγοι βέβαια νέοι εκλέγονται σε θέσεις σημαντικές. 1,6% των ευρωβουλευτών είναι νεότεροι των 29 ετών. Δεν εκφρα... Ε, αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται στο πολιτικό σύστημα οι νέοι, πράγμα το οποίο ξάνει και τη δυσπιστία τους στο μέλλον. Δεν είναι ανόητοι οι νέοι. Εάν δουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι παράλογο, δεν θα συνεισφέρουν στην ε, συνέχιση του. Όταν ακούνε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο για τους πολιτικούς που είναι διεφθαρμένοι, σταματούν να ψηφίζουν και αρχίζουν να συμμετέχουν με άλλους τρόπους εκτός από τις ε, ε, δομές. Όταν μαθαίνουν ο μόνος τρόπος να βρουν δουλειά είναι να είναι από την κατάλληλη οικογένεια, να ξέρουν τον κατάλληλο ε, άτομο και να είναι μέρος του συστήματος αντιδρούν. Το έρασμος είναι ένα πρόγραμμα που θέλει να ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα ε, των νέων στην Ευρώπη. Εγώ για έξι μήνες παρακολούθησα τα προγράμματα Erasmus και κατά διάρκεια αυτού του εξαμήνου υπήρχαν τόσο πολλά σκάνδαλα μεταξύ των πολιτικών που πραγματικά και εγώ που είμαι προευρωπαία, σε να διαρωτώ με, είναι ε, τα πράγματα και πάρα πολλά προβλήματα υπήρχαν και μεταξύ των νέων της χώρας την οποία τώρα, της Πορτογαλίας. Και δεν πρόκειται για προβλήματα που αντιμετωπίζουν μόνο οι νέοι στην Πορτογαλία και αλλού τα αντιμετωπίζουν. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι τόσο βρεστά έπρεπε πράγμα το οποίο είναι απογοητευτικό. Ποτέ δεν ήταν ε, τόσο ενεργή πολιτικά η νέα ε, όσο σήμερα μόνο οι συγκρίσει με το πριν από 50 χρόνια και τι γινόταν οι ίδιε χώρε θα μπορούσαν να μα δίνουν στρατικά αποτελέσματα. Παρά το γεγονό όμω ότι δεν ψηφίζουν οι νέοι, έχουν μεγάλη συμμετοχή σε κινήματα στην κοινωνία των πολιτικών, συζητούν στο ίντερνετ και όπου μπορούν για τα προβλήματα πολιτικά. Τους ενδιαφέρουν όλα τα προβλήματα περιβαλλοντικά, το προσφυγικό κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα και χωρίς τα νέοι θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος και την παρχουσών δομών. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και τα επόμενα 20 χρόνια δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολιτικοί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η δημοκρατία είναι μια συνεχής και επίπονη δουλειά μεταξύ όλων των γενεών ώστε να υπάρχει συμμετοχή δημοκρατική των πάντων. Δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιέστε. Έχουμε εταιρική σχέση μεταξύ των σχολείων και των οργανώσεων των νέων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οπότε έχουμε αυτή η διαμόρφωση τη πολιτική μια συμμετοχή. Και επομένω νομίζουμε θα πρέπει το όριο να είναι τα 16 και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μην έχουμε πολιτικού φραγμού και να είναι ευκολότερο το να ψηφίσει κανεί και ακριβώ όπω είπαμε να έχουμε και την ηλεκτρονική ψηφοφορία και να έχουμε εκλογικά κέντρα σε σχολεία, σε σε, σε, σε βιβλιοθήκες αυτό με τη γραφή στους καταλόγους και περισσότερη ευελιξία αν κανείς δεν κατοικεί στον ε, τόπο ε, όπου έχει καταχωρηθεί. Οπότε θα πρέπει έτσι να εμπλακούν οι νέοι στην ε, λήψη των αποφάσεων και αυτό θα γίνει αν τους αφήσουμε να επηρεάζουν όλα αυτά που αφορούν τη ζωή τους και αυτό ε, θα μπορούσε να έχει διαρκή χαρακτήρα και θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδου ε, δομέ και οι νέοι να επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων και έτσι σε, ένα, ε, σε μια περίοδο 10 ετών από τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε την πραγματική δημοκρατία. Αλλά τελευταίο και σημαντικό έχουμε την κοινωνία των πολιτών, έχουμε ισχυρέ οργανώσει τη νεολαία και ε, εκεί ε, αποκτούν τις δεξιότητες, εκεί μαθαίνουν πώς γίνονται οι προεκλογικές εκστρατείες, πώς γίνονται οι συζητήσεις, οι από ε, το θεμέλιο της δημοκρατίας και δεν είναι πυρηνική δυσική όλα αυτά και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που τηρήσατε τον ε, χρόνο της ακρόασης και πάμε τώρα σε την τελευταία ομιλήτρια που είναι η κυρία Αντριάννα Κος η οποία έχει ήδη υποβάλει κάποια αναφορά και είναι μια αναφορά που αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι η αναφορά 2651 του 14. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό αφορά το θέμα μας ε, και από ό,τι κατάλαβα εδώ πήγε καλά η αναφορά, δεν είναι ένα θέμα όμως τόσο αγαπημένο του Συμβουλίου. Τέλος πάντων, κυρία έχετε τον λόγο. Ε, γεια σας, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η κυρία Κος. Σας ευχαριστώ γιατί έτσι κατέστη δυνατόν να εξηγήσω την αναφορά που αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είμαι ε, Σλοβένα, νέα ε, Σλοβένα και έχω μελετήσει μία σειρά αναφορών. Έχουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Ε, να σας πω στο τέλος ποια είναι τα συμπεράσματά μου. Αυτό το οποίο πρότεινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήταν μια αναφορά την οποία συνέταξαν φοιτητέ. Ε, αφορούσε κάποιους ε, αφορούσε εκλογές ε, για το Ευρωκοινοβούλιο. Και είπαμε για πώς θα καταφέρουμε να ελκύσουμε περισσότερους νέους να ψηφίσουν. Γιατί στην Σλοβενία έχουμε μεγάλη αποχή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στην Σλοβενία ε, είναι μια πρόταση που ανάγεται στο 2003. Αυτό το πρότειναν Σλοβαίνοι Ευρωβουλευτές. Όμως η ιδέα αυτή δεν έπιασε τόπο. Έχουμε τώρα τις εξής απόψεις. Έχουμε ψηφοφορία, i-voting και e-voting. E-voting σημαίνει ψήφιση με ε, ηλεκτρονικές συσκευές και i-voting γίνεται με υπολογιστή. Και αυτό αφορά και την περισλογή των ψήφων για μας ευμένως. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την ιστοσελίδα που θα ε, βοηθά στη λειτουργία του το iVoting. Άρα θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κάποιους κανόνες, κάποιο πλαίσιο, κάποιες προθεσμίες. Και έτσι αυτή η ιδέα να υλοποιηθεί. Επίσης, θέλουμε να καλύψουμε και τους ευρωβουλευτές. Δηλαδή, έτσι ο κόσμος να έχει το περιθώριο να εξοικειωθεί με αυτούς τους νέους τρόπους ψηφοφορίας. Αυτό βέβαια να γίνει βαθμία. Και υποβάλαμε το 2014 αυτήν την αναφορά όπως αναφέρατε πρόεδρε. Από τότε ε, εστιάστηκε η προσοχή μας βέβαια ε, στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Πάντως εγώ θεωρώ ότι το e-voting, η ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, θα κρατηθεί στην επικαιρότητα μια που η τεχνολογία προχωρεί με άλματα. Ε, και το διαδίκτυο βεβαίως πάντα θα βοηθεί, οπότε ε, θα βγει από το ψυγείο ούτως επίν αυτή μας η ιδέα. Οπότε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, το e-voting, ε, θα μπορέσει ο ψηφοφόρος να ψηφίσει όπου και να βρίσκεται. Είτε στη χώρα του είτε στο εξωτερικό. Και έτσι θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση ε, σε μια ενημέρωση. Θα υπάρχει μέσα μια διαδικτυακή πύλη το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για την ασφάλεια του συστήματος. Το 2014, τον Μάιο, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο και αναφέρεται εκεί ότι στην Εστονία έγινε μια δοκιμή ηλεκτρονική ψηφοφορίας. Το συμπέρασμα ήταν ότι το σύστημα δεν ήταν στεγανό από πλευρά ασφάλεια και ότι δεν μπορούσαν να εξαπολυθούν κυβερνοεπιθέσεις προς το σύστημα. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν φταίει το σύστημα κατά τη γνώμη μου ε, ήταν ε, πρόβλημα εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων εκείνων δηλαδή που θα όφυλαν να χρησιμοποιήσουν και όχι να καταχραστούν του συστήματος. Η πολιτική ε, έχει κατά κάποιο τρόπο υποβαθμιστεί, έχει χάσει αξιοπιστία, έχουμε σκάνδαλα, έχουμε διαφθορά, ε, νομίζω ότι τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα, θα βοηθηθεί η πολιτική με την λειτουργία ψηφοφορία. Δεν μιλούμε για κανένα μαγικό ραβδάκι, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Ίσως βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σήμερα και άρα θα πρέπει να λάβουμε κάποιες κρίσιμες αποφάσεις. Και να σας πω κάτι το το έλεγε ο Καρλ Ρέμψ. Αυτός είχε εφεύρει μια συσκευή και για τις εφευρίες του έψαχνε επενδυτή. Οπότε δεν, κανείς δεν του δάνειζε χρήματα και του λέγανε ότι ε, και, να, ε, δεν σας δίνουμε χρήματα, έχουμε άλλο. Είδατε όμως η τεχνολογία που μας οδήγησε. Ευχαριστούμε και τώρα εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αγορητών, των προσκεκλημένων μας στον πάνελ και τώρα πέστε μου ποιος θέλει το λόγο, κανείς μας δεν ζητήσει το λόγο. Όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει το λόγο, πάντως σε 25 λεπτά θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Κυρία Σπινέλη είναι η πρώτη που ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όσον αφορά την κρίση που περνά η δημοκρατία, κάτι για το οποίο ακούσαμε, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι το τι λένε ε, τα κινήματα διαμαρτυρίας σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λένε και οι εθνικιστές αυτοί που μάχονται για την εθνική κυριαρχία που πολλές φορές διακρίνονται από ξενοφοβία. Τι μας λένε. Μας λένε πρώτα πρώτα ότι έχει ξεπεραστεί ε, ο θεσμός του κόμματος και ότι θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι συμμετοχής. Νέοι τρόποι συμμετοχής που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται. Κάτι άλλο το οποίο μας λένε αυτοί οι επικριτές είναι το ότι η αποχή μειώνεται λόγω αυτών των κινημάτων. Άρα, να το είδα στη Γερμανία, ξέρετε, ή στις ε, εκλογές του Σαββατοκύριακου, τις περιφερειακές. Έχει ξανατονωθεί η πολιτικοποίηση στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και δεν συμφωνώ με την πρόταση τη σχετική με την αποχή στις ευρωεκλογές. Ότι δηλαδή δεν είναι πρόβλημα, όπως μας είπε ο δόκτωρ Μπερτοντσίνη. Και ότι όποτε παρεμβαίνει το κράτος δεν έχουμε ε, χωρίς την παρέμβαση του κράτους τέλο πάντων ικανή συμμετοχή. και τα συμπεράσματα τα οποία μπορώ να εξαγαγώ είναι τα εξή. Ότι υπάρχουν κάποιες υπερκρατικές, υπερεθνικές οντότητες και πλατφόρμες όπως ανέφερε ο κύριος Νταφ. Πολύ σημαντικές. Αλλά θα πρέπει τώρα να δούμε ποιες είναι οι βασικές θεματικές ενότητες για τις οποίες θα μπορούσε να γίνει κάποιο ε, είδους ε, τέτοια συσπήρωση υπέρ εθνικές ε, το να ενισχύσουμε οικονομικά τα υπάρχοντα κόμματα να έχουμε κάποιον αλλοδαπός υποψήφιο σε εθνικές εκλογές είναι τώρα αυτά θέματα τεχνικά, τεχνοκρατικά. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις και κάτι που ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή είναι το εξή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ε, ισχυρό εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου. Σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν ευρωπαϊκές επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές είναι αυτές που δικαιούνται να προετοιμάζουν τέτοιες συναντήσεις. Αν λειτουργούν σωστά, οι εθνικοί βουλευτές μπορούν μέσω των εθνικών αυτών επιτροπών να προετοιμάσουν τις συζητήσεις με τους υπουργούς και έτσι μπορούν να προετοιμάσουν πραγματικά με συμμετοχή πολλά ζητήματα. Σίγουρα αυτό προαπαιτεί μεγάλο όγκο δουλειά. Δεν γίνεται με το τίποτα, αλλά θα βοηθούσε για να νομιμοποιήσει πολύ πιο πολύ το έργο των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα προτίμαζα και τους υπουργούς, γιατί και αυτοί θα έρχοντουσαν καλά προετοιμασμένοι για να συμμετέχουν στις συζητήσεις με τα άλλα κρατημέλη. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικό, πραγματικά να σας υπογραμμίσω την δυνατότητα αυτή. Στη Δανία την πατρίδα μου ήμασταν αυτοί που το περάσαμε το 1993. ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά για να το θέσουμε ευγενικά. We don't see the names, we don't, so somebody... ονόματά σας, βλέπω κάποιον εκεί πίσω που θέλει το λόγο. Μας πείτε ποιος είστε. Είμαι ο Λουίς Φερνάντε. Είμαι Ευρωπαίος πολίτης. Και παίρνω το λόγο γιατί σήμερα μιλούμε και σας ευχαριστώ που έχετε οργανώσει αυτή την ακρόαση για την Ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η ηθαγένεια, η κοινοτική, θεωρητικά είναι κάτι που στήσεται στην ηθαγένεια του καθενός, αλλά είναι κάτι το οποίο πολλές φορές ε, έχει προβλήματα και υφίσταται κάποια εμπόδια. Βλέπουμε και πολίτες ε, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που παίρνουν κάποιες αποφάσεις που είναι κατά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και κατά της ε, Ευρωπαϊκής Ιθογένειας. Ως Ευρωπαίος πολίτης, παρά το γεγονό ότι δεν είμαι μέλος αυτών των χωρών, πιστεύω ότι με αυτή την έννοια και τα δικαιώματα μειώνονται. 10 με 11 χρόνια πριν κάναμε στην οργάνωση του Μια εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Και ο τίτλος ήταν «Ψηφίστε, είναι το δικαίωμά σας». Δεν ήταν όμως το δικαίωμα όλων των ανθρώπων που ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ. Υπέρ, ναι, ψήφισαν οι περισσότεροι πολίτες σε όλες τις χώρες. Δύο κράτη-μέλη δεν ψήφισαν και οι πολίτες αυτών των δύο χωρών επηρέασαν τα δικαιώματα όλων των άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Εάν λοιπόν δεν δώσουμε μια θετική απάντηση σε όλα τα άτομα τα οποία πιστεύουν ότι το ευρωπαϊκό όνειρο, αν θέλετε, πλέον δεν είναι πραγματικό δεν αντιποκρίνεται τι προσδοκίες τους, δεν θα κάνουμε τίποτε. Ο κύριος Νέμι μίλησε για το μεγάλο, τη μεγάλη δημοκρατική πρόκληση, αν θέλετε, και πώς θα την υλοποιήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε πρώτα απ' όλα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίζουν σε οτιδήποτε άπτεται κάτι του Ευρωπαϊκού και του αφορά, όπου και αν βρίσκονται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Σύντομα παρακαλώ για να μπορέσουν να απαντήσουν και ομιλητές. Γεια σας, το όνομά μου είναι Χέμα Μαρτίνεφ. Εμείς ε, συμμετείχαμε στην δημόσια ε, διαβούλευση επιτροπής. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε δημοκρατική υποστήριξη. Μιλάμε για θέματα ενδιαφέροντα όπως είναι η κοινότητα, η, δημοκρατική συμμετοχή και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Οι Ευρωπαίοι έχουμε λίγε δυνατότητε να συμμετέχουμε στι δημοκρατικέ διαδικασίε. μόνο μέσα τη ψηφοφορία τη ευρωπαϊκής και δύσκολα μπορούμε να πείσουμε του συμπολίτε μα να ψηφίσουν. Αν όμως, επιπροσθέτως υπάρχουν και εσωτερικές δυσκολίες για να ψηφίσει κάποιος, τα πράγματα γίνονται αδύνατα. Θα ήθελα να δώσω το παράδειγμα της χώρας μου. Το 2011, σύμφωνα με την εκλογική μεταρρύθμιση, για όλους τους Ισπανούς που ζούμε στο εξωτερικό, 2 εκατομμύρια περίπου, το να μπορέσουμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Στις τελευταίες ευρωεκλογές λιγότερο του 2% των ε, Ισπανών που ζούμε εκτός Ισπανίας μπορέσαμε να ψηφίσουμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πραγματικά υπάρχει ένα συμπληρωματικό πρόβλημα που προστίθεται στην απογοήτευση από την Ευρώπη. Ποτέ δεν ήταν πολιτικοποιημένα τα πράγματα και οι άνθρωποι που σήμερα και οι Ισπανοί θέλουν να συμμετάσχουν στο γίγνεσθε της Ευρώπης. Στις ε, τελευταίες μας εθνικές εκλογές, τις βουλευτικές, τον Δεκέμβριο, μόνο μπορέσαμε να ψηφίσουμε 100.000 Ισπανίοι που βρίσκονται εκτός Ισπανίας. 5% μόνο. Απλώ ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός και να ζητήσω στους ευρωπαϊκούς δεσμούς να επαγρυπνούν ώστε στις διάφορες χώρες να δοθεί η δυνατότητα ίση όρη να επιτρέπουν στους πολίτες τους αν βρίσκονται να μπορούν να ψηφίζουν. Παρακαλώ. Είμαι ο Τζέριλ Κρίστον Χάνκελ, είμαι Γερμανό και με τον δόκτωρο Φρονσό Μενεγάλ είμαι συμπρόεδρος και συνειδητής του EuroSoc, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή σε ε, νόμιμο ε, καθεστώτος ευρωπαϊκού χωρί ε, ε, μη κερδοσκοπική. Ε, πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Κύριε Νίμης, Το καθεστώς μιας, ενός ευρωπαϊκού σωματείου είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες. Οι ευρωπαϊκοί πολίτες μπορούν μόνο να οργανώνονται μόνο σύμφωνα με την, ε, ε, τα ισχύοντα στην νομοθεσία, στην εθνική τους νομοθεσία και όχι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο. Είχα μια συνομιλία με τον κύριο Μάρτιν Ζενμάιερ, πεύθυνο του γραφείου του πρόεδρου Γιούνκερ και μου είπαν ότι αυτή η επιτροπή δεν θα αναλάβει να κάνει τίποτα για την επίλυση του θέματος. Αλλά στα πλαίσια των 10 προτεραιοτήτων του πρόεδρου Γιούνκερ, στο σημείο 10 ανέφερε ο πρόεδρος και ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να προωθήσει και την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα κάνει τίποτε επί αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος εδώ. Έχω μια ερώτηση για το δικαίωμα πρωτοβουλίας. και προς τα μέλη του πάνελ. Ποια είναι η απόψή σας Εάν επιτρέπουμε σε κάποια άτομα να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις για θέματα νομοθετικά δεν σημαίνει ότι εκείνοι θα κάνουν την νομοθεσία. Ίσως αυτό που λένε είναι να βοηθήσουν τους, νομοθέτου, τους νομοθέτες να τους δώσουν κάποιες ε, καινούργιες ιδέες. Εάν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν, τι έχετε να προτείνετε στα πλαίσια του, ε, της δικιά μας πρωτοβουλίας αυτού που υπάρχει. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τζένκη. Θα σας τα πω τηλεγραφικά. Το πρόβλημα της αποχής των νέων από τις εκλογέ είναι σίγουρο πολύ σημαντικό και πιστεύω συμφωνώντας με την κυρία Σπινέλη όσον αφορά τις λύσεις που δεν μπορεί να είναι τεχνοκρατικού χαρακτήρα αλλά κοινωνικού δηλαδή να σταματήσουν οι φραγμοί που υπάρχουν με κάποια επικοινωνία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακριβώς όπως ε, αναφέρθηκε. Μια τέτοια λύση ε, πρέπει να συζητηθεί. και δεν θα πρέπει να κολλάμε στο θέμα της ε, ασφάλειας για αυτές τις πιθανές ε, λύσεις. Θα μπορούσε να υπάρχει κρυπτογράφηση, θα μπορούσε να υπάρχουν κάποιες ψηφιακές υπογραφές και άλλος τρόπος ε, ταυτοποίησης ψηφιακής. Και έτσι μπορεί να υπάρχει ακόμα και διπλή κρυπτογράφηση. Επομένως θα πρέπει στα σοβαρά να αναπτυχθεί μια προβληματική ούτω ώστε να πέσουν αυτοί οι φραγμοί. Είναι κοινωνικό το θέμα, όχι οικονομικό και να μην υπάρχει αυτή η απομόνωση μεταξύ των νέων και του σκοπού, α το πούμε, του τελικού που είναι το να γίνουν οι εκλογές. Κύριε Νέμιτσα, αρχίστε εσείς, είχατε και εσείς ερωτήσεις που σας υπευλήθησαν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να σας πω δύο λόγια. Να, εδώ από δεξιά, δηλαδή ότι έχουμε την εντοπιστική δημοκρατία και την άμεση δημοκρατία από την άλλη μεριά και δεν θεωρώ ότι μία είναι χειρότερη από την άλλη. Έχουμε στην Ευρώπη τώρα αντιπροσπευτική δημοκρατία και δεν αποκλεί την συμμετοχική δημοκρατία. Αλλά η ουσία δεν είναι το να πηγαίνει ο κόσμο να ψηφίσει, έτσι και του ψηφίσει σε μια δημοκρατία. Το θέμα κανεί να εμπλέκεται για να μπορεί έτσι να επηρεάσει και πέραν τη ψήφου και των εκλογών. Αυτό είναι το αφήγημά μας και αυτό σημαίνει ότι κανείς αλλάζει τα πράγματα προς το καλύτερο αντί να λέει κούφια λόγια για νόμους και διατάξεις. Αυτό θα πρέπει να γίνεται επομένω τη σημερινή μέρα. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση και ο κόσμος έτσι αλλάζει και όχι με το να πετάει βόμβες μολότοφ στα σπίτια όπου καταλύουν οι αιτούντες άσυλο. Επομένως έτσι θα πρέπει με τον φυσιολογικό τρόπο να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο από εδώ, από τις Βρυξέλλες. Για την πρωτοβουλία, ναι θέλουμε να υπάρχει παντού εμπλοκή του κόσμου, θέλουμε να εστιάσουμε προσοχή μας στα πολιτικά κόμματα, γιατί λένε στα κρατημέλη ότι μόνο οι πολίτες κάποιας χώρας μπορούν να είναι μέλη ενός κόμματος ή να φτιάξουν ένα κόμμα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει πολλά πράγματα παρά το αυτό που ελέγχθη. Μπορεί να μην το λέει το πρόγραμμα εργασίας. αυτό το σημείο ότι έχετε καλέ ιδέες. Οπότε να μου τις πείτε και θα τις ε, λάβουμε υπόψη. Κάνουμε ό,τι περνάμε το χέρι μας τόσο να θέλουμε τους νέους να μπλακούν στο παιχνίδι τη δημοκρατία Τώρα, για την... τις εθνικές ψηφοφορίες, τις εθνικές εκλογές. Και τι κάνουν στις εθνικές εκλογές αυτοί που έχουν φύγει από τη χώρα. Κάποιοι λένε ότι κάποιο θα πρέπει να ψηφίζει εκεί που κατοικεί. Αυτό είναι μια σχολή σκέψης. Αυτό γίνεται το ίδιο σε επίπεδο τοπικών εκλογών και ευρωεκλογών. Κάθε νέας μπορεί να ψηφίσει εκεί που κατοικεί. Υπάρχει μας και άλλη σχολή σκέψη, άλλη άποψη. Θα πρέπει ακόμα και κανείς έχει αποδημήσει να μπορεί να ψηφίσει την πατρίδα του. Στη συνθήκη προβλέπεται ότι ο κόσμος ψηφίζει εκεί όπου κατοικεί. Να, επομένως, οι νομικοί βάσει να εξαναγκαστούν τα κράτη-μέλη να δεχθούν ότι εκείνοι που έφυγαν από τη χώρα μπορούν να ψηφίσουν στην πατρίδα τους. Βέβαια δεν νομίζω, δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι αν αυτό είναι νομικά εφικτό. Δεν ξέρω, για την πατρίδα μου αμφιβάλλω πολύ. Γιολάινεν, θέλετε να μας πείτε κι εσείς. Ναι, να καλάσουμε τη νέα γενιά να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Δημοκρασία και στις ευρωεκλογέ. Και γι' αυτό, Ντανούτα, προτείναμε να μειωθεί το όριο ηλικία για την ψηφοφορία στα 16 χρόνια. Το έχει κάνει αυτό η Αυστρία και επίση να εισαχθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεύτερο θέμα, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση γιατί λείπουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το είπε και η συνάδελφο. Οτιδήποτε λοιπόν θα μπορούσε να ενισχύσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ ομάδε στι συζητήσει και στην προεκλογική εκστρατεία θα ήταν ωφέλιμο και ακρογωνιαίος Λίθος θα είναι οι ευρωπαϊκές λίστες. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε και με τον Σπίτιν καντιντάτ, με τον ε, κορυφαίο αυτόν υποψήφιο. Προς τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, να το πω το εξής, να προσέξουμε, να προσέξουμε γιατί δεν θα πρέπει να αντιπαραθέσουμε και να αντιδιαστέλουμε την ε, ευρωπαϊκή με την εθνική υπηκότητα. Γίνονται όλο και πιο πολλά ευρωπαϊκά, εθνικά μάλλον δημοψήφισματα για ευρωπαϊκά ζητήματα. Είμαστε μια κοινότητα 28. Ακόμα και να έχει αποφασίσει και έχει αποφανθεί λοιπόν ένα κράτος παραμένουν και άλλα 27. Είναι λίγο... Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, γιατί και στα κοινοβούλια ακόμα το ακούμε ότι «Μα αυτό είναι η δημοκρατία». Ναι, η δημοκρατία είναι, αλλά ελοχεύει και ένα κίνδυνος σοβαρός. Α κοιτάξουμε τα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα. Γιατί όχι αν θέλουμε άμεση δημοκρατία για ευρωπαϊκά ζητήματα. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σοπλίν. Ευχαριστώ για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Νομίζω τα πράγματα είναι και τα προφανή. Δεύτερο θέμα για τον κύριο Νέμιτ. Πολλοί ακαδημαϊκοί διατείνονται ότι η ανακατανομή της εξουσίας προς την κοινωνία των πολιτών, τα λόμπι, τη ΜΚΙΟ, ε, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου. Όλοι πιστεύουμε λοιπόν ότι καλή είναι η κοινωνία των πολιτών, αλλά είναι σαφής ε, η τάση τα τελευταία 56 χρόνια. Μία ερώτηση τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα πίσω έδρανα. Έξω, όσων καταλαβαίνω υπάρχουν ευρωπαϊκές αρχές, ε, ευρωπαϊκές αξίες οι οποίες είναι γραμμένες στην πέτρα. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Θα πρέπει και να υπάρχει και σκεπτικισμός αν θέλετε. Η δημοκρατία προϋποθέτει ότι ακούμε όλες τις τοποθετήσει, τις κριτικές, τις αξίες όλων των πολιτών, είτε είμαστε υπέρ είτε κατά. Αν τα αρνηθούμε αυτά, πώς θα δεχτούμε όλους τους πολίτες. Και τελευταίο θέμα για την νεολαία. Ναι, αλλά να θυμόμαστε ότι τα άτομα τα οποία είναι τώρα 20-30 χρονών θα φτάσουν 120-130 χρονών ενδεχομένω με την τεχνολογία. Άρα υπάρχει μεγάλη τάση προς πιο μεγάλες ηλικίε. Και θα είμαστε νεότατοι στο μέλλον εμείς οι 65 Ο Άντριου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συνθήκη στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ περιοριστική. Περιορίζει πάρα πολύ το τι μπορεί να πετύχει κανείς ως βελτίωση της ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ελπίζω το Κοινοβούλιο κατά την προετοιμασία του πακέτου για την επόμενη συνθήκη θα συμπεριλάβει και μία αναθεώρηση του άρθρου 22 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά και τα δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά ζητήματα Και ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χαλαρώσει επίσης και τις περιορισμούς για τους σκοπούς ε, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Ότι πρέπει να πρόκειται δηλαδή για νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό είναι παράλογο. Και πάντα πίστευα ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών θα έπρεπε να αποτελεί ένα μέσο κίνησης, αν θέλετε, στο οποίο θα αναγκάζει τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν τις γενικότερες εκστρατείες πολιτικής μεταρρύθμισης για τη διαδικασία ελέγχου των εθνικών κοινοβουλίων. Συμφωνώ, συμφωνώ. με την κυρία συνάδελφο ότι η εμπειρία μας ε, από τις σκανδιναβικές κυρίως χώρες είναι χρήσιμη. Αλλά το να δώσουμε υπερβολικό βάρος στις εθνικές ε, ανησυχίες, όπως είδαμε για παράδειγμα και στη Βρετανική περίπτωση για την απόφαση της 19ης Φεβρουαρίου, όπου το Συμβούλιο παραλόγως πως αποφάσισε να υπάρξει με τέτοια κόκκινη κάρτα. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια λανθασμένη κατεύθυνση. το μηχανισμό έγκυρης προειδοποίησης, για παράδειγμα, θα τον καταργούσα. Θα επέτρεπα στα εθνικά κοινέμβουλια να αποφαίνονται για όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα, σε όλα τα επίπεδα της νομοθετικής διαδικασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σόρενσεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να αντιδράσω στα διάφορα τα οποία ελέγχθησαν για την συμμετοχή στην πληροφορία των νέων. Συμφωνώ ότι η συμμετοχική δημοκρατία ξεπερνά το να πάει κανείς και να ψηφίσει μόνο μια μέρα. Δεν είναι θέμα ε, τεχνικών προσαρμογιών για να αυξηθεί το ποσοστό των νέων που ψηφίζουν. Τα ε, μέσα δικτύωσης είναι επίσης ε, ε, μέσον, μέρος της λύσης. Και τι θέλω να πούμε στους πολιτικούς. Ας δούμε στα κοινωνικά δίκτυα πόσες αντιδράσεις υπάρχουν, πόσοι για σας τους πολιτικούς έχουν να πούν κάτι το θετικό ή όχι. Δεν μπορούμε για τους νέους ε, να μην ε, διασυνδέουμε τις δομές με τις αποφάσεις και τις δράσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε όλοι πώς μπορούμε να προκαλέσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων για το γίνεται στην πολιτική. Βεβαίως και υπάρχουν και τεχνικές ε, λύσεις αν θέλετε για να αυξηθεί η συμμετοχή τους. Στην Δανία έχουμε και ε, κάλπες για να ψηφίζουν οι νέοι και σε βιβλιοθήκες και εκεί που βρίσκονται οι νέοι. Τους στέλνουμε μηνύματα για να τους υπενθυμίσουμε ότι γίνονται εκλογές σε δύο μέρες. Και τους υπενθυμίζουμε κάποιες ε, λεπτομέρειες και όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα είδαμε ότι αύξησαν τη συμμετοχή των νέων. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό δεν είναι να βάλει τα βρουλάκια κάπου ο νέος. Είναι όταν ε, έχουν πρόσβαση στην ψηφοφορία πρέπει να δούμε ότι θέλουν και πληροφορίες άλλες και θέλουν να ξέρουν γιατί ψηφίζουν από τεχνικής πλευράς μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να γίνει πιο προσβάσιμη η ψηφοφορία θέλει στους νέους. Διότι θέλουν ενημέρωση και ενδιαφέρονται για τα συζητήσεις που γίνονται και σε πολιτικό επίπεδο γιατί τους ενδιαφέρει το πολιτικό ε, γίγνεσθε. Μία συγκεκριμένη ερώτηση έγινε από τον νεαρό που αφορά την, ε, το δικαίωμα ε, της... Ε, πρωτοβουλίες και το ευρωπαϊκό αυτό δικαίωμα. Δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Έτσι προβλέπεται στην συνθήκη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε να κάνει μία νομοθετική πρόταση επί αυτού του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικαίωμα λοιπόν πρωτοβουλίας προς το παρόν αυτά μας επιτρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία ε, οι δύο συνομοθέτες έχουν αποφασίσει. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν ενδιασμοί εκ μέρους των πολιτών όταν πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιου πρωτοβουλίες όπως ελέγχθη να δίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ταυτότητά τους. Υπάρχουν ενδιασμοί και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της ε, εφαρμογής του ECI, αυτή του δικαιώματος πρωτοβουλίας. Δεδομένου ότι πολλές φορές ε, τα... είναι πολύ πλοκό το θέμα του τι είδους δεδομένα θα στείλει κάποιος και κυρίως όσον αφορά την συμμετοχή του σε κάτι το οποίο είναι μόνο μία πρωτοβουλία. Ε, Γιώζεπ, Τελειώσαμε, εσύ δεν θέλεις το λόγο και θα ήθελα να ενθαρρύνω τους πάντες, αφού τους ευχαριστήσω, να παραμείνουν και το επόμενο θέμα μας, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό. Thank you very much for leaving those who live. Thank you very much for staying. Θα θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που θα φύγουν από την αίθουσα και να ευχαριστήσω και αυτούς που θα παραμείνουν στην αίθουσα. Reaction. Sorry. yeah. Thank you. Uh, those who leave, thank you very much for leaving. Thank... Λαμβάνει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ όσους φεύγουν και ευχαριστώ και όσους μένουν. Ευχαριστώ τους πάντες δηλαδή. Τέλεια. That's really perfect. Thank you. But do it, please. So, we'll start. Thanks. Θα αρχίσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα το τελευταίο πάνελ μας. Τα δικαιώματα των πολιτών απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κύρια θέματα που είναι δύο θα είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς θα ε, μπορέσουμε να κάνουμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ε, την ε, αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε λειτουργικό επίπεδο και μετά ε, και πώς θα μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερο στην ε, πολιτικές που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο είναι το δικαίωμα αναφορών. Πρώτα απ' όλα δίδω το λόγο συνάδελφό μου κυρία Τζουντ Κίρτον Ντάρλινγκ. Αρχίζοντας θα ήθελα να σας πω ποια είμαι και τι έχω κάνει. Διότι οι ομιλητές σήμερα στην ακρόαση, από την άποψή μου, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ ήμουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο το, από το Μάιο του 2014 και πριν εκλεγώ εδώ ήμουν εκλεγμένη συγκαλιστική εκπρόσωπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάρα πολλά χρόνια πρέπει να πω ότι υπερασπίστηκα τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων εργαζομένων και των πολιτών της Ευρώπης εκτός ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και τώρα είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών. Είμαι λοιπόν σε μια διαφορετική θέση και ακούω τους πολίτες να μιλούν για προβλήματα τα οποία έχουν με την Ευρώπη και έρχονται εδώ οι αναφορές τους στην Επιτροπή Αναφορών και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία που έχω από το Μάιο του 2014 και μετά από την αντίπερα όχθη. Είναι λοιπόν προνόμιο για μένα να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, γιατί πιστεύω βασικά ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την αυξημένη δημοκρατική συμμετοχή στους χώρους εργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εργασιακά δικαιώματα, συνδικαλιστικό επίπεδο, σε κοινοβουλευτική δημοκρατία και σε αυξημένες εξουσίες που θα δοθούν για την δημοκρατική διακυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δημοκρατικό δικαίωμα που έχουν όλοι οι πολίτες να κάνουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αγωνίζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των. Οι δραστηριότητες της Επιτροπής μας ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής και είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι είναι το μόνο μέρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο ως Επιτροπή έχουμε ημερήσια διάταξη που καθορίζεται πλήρως από τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών και από τα θέματα τα οποία τίθενται, είμαστε κατά κάποιο τρόπο η γέφυρα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Και είναι ίσως ένας από τους καλύτερους τρόπους του οποίου μπορούν να απευθύνουν άμεσα και απευθεία ε, ε, τα αιτήματά τους, τις ανησυχίες τους ε, και τις έγνοιε τους στου ευρωπαϊκούς θεσμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε σημαντικοί. Και βεβαίω, αν μπορούσα να εκφραστώ ως ε, Ευρωβουλευτή θα έλεγα με κάπω πιο επικριτικό πράγμα ότι δεν πρέπει ε, πνεύμα ότι κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν καταλάβει το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών και πολλές φορές ε, τίθεται ένα αμφιβόλο τρόπος που λειτουργούμε και εμείς και τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να πω ότι το 2009 έλαβε η Επιτροπή μας 2.000 αναφορές, το 2014 3.000. Αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός τους και βεβαίως όλες περνούν από ένα φίλτρο για να δούμε αν είναι παραδεκτές, ε, ε, αν, είναι, αφορούν θέματα τα οποία άπτονται των κοινοτικών ε, θεμάτων και πρέπει να πω από τις 3.000 χίλιες και μπορούσαν ε, θεωρήθηκαν ε, ε, παραδεκτές και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε σχεδόν όλες οι αναφορές να γίνουν παραδεκτές παρά τη γνώση ότι μερικές είναι κάπως ιδιότυπες. Ο κύριος όγκος των αναφορών αυτών τι σημαίνει ότι υπάρχει γενικότερα μία πίεση που ασκείται σε όλους μας ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά και λειτουργούμε και να δώσουμε αποτελεσματικές και ταχύες λύσεις. Η ποικιλία των θεμάτων που περιέχονται ε, στις αναφορές σημαίνει ότι εμείς οι Ευρω... οι Ευρωπαίοι, ε, οι, Ευρωβουλευτές γινόμαστε εμπειρογνώμονες επί παντός του πιστητού όπως τα λέγαμε για να μπορέσει κανείς να ε, ασχοληθεί με το σύνολο των προβλημάτων που μας υποβάλλονται θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα από τεχνικής πλευράς και από οποιαδήποτε πλευρά. Πιστεύω ότι κάνουμε σχετικά καλά τη δουλειά μας. Πάντα βεβαίως όλα είναι τελειοποιήσατε, αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξη. Το βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι και απογοητεύομαι πολλές φορές στην ε, Επιτροπή μας από τη στάση κάποιων κρατών μελών προς τους πολίτες ε, οι οποίοι μας υποβάλλουν τις αναφορές τους. Ένα παράδειγμα, όταν γίνεται λόγος για το δικαίωμα ψήφου και αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ. Όταν τίθενται τέτοιου είδου θέματα για τους εκπατρισμένους του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν ζουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνησή μας ε, είχε πει ότι τέτοιου είδους δικαίωμα θα δοθεί σε όλους τους ε, εκπατριστέντες με θετικό πνεύμα το αντιμετώπισαν, αλλά τελικά δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Τώρα θα έχουμε το δημοψήφισμα σε λίγους μήνες. Και βεβαίως πρόκειται για σημαντική απόφαση για τη ζωή μας και οι Βρετανοί που ζουν στο εξωτερικό δεν έχουν λόγο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως απογοητευτικό και πολλές φορές όταν τίθενται τέτοιου είδους θέματα δεν έχουμε και την κατάλληλη υποστήριξη στα κράτη-μέλη για να την υποστηρίξουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχει με το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή πάρα πολύ καλή συνεργασία εκ μέρους μας. Κάποιος από το γραφείο του Διαμεσολαβητή επίσης ε, θα πάρει το λόγο. Πρέπει να πω ότι επίσης με θέματα που αφορούν ε, τους ε, μετανάστες, τους πρόσφυγες, είδαμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων. Μόνον έτσι μπορεί να ακουστεί περισσότερο η φωνή του κάθε Ευρωπαίου πολίτη που επηρεάζεται από τέτοιου είδους θέματα και να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Ίσως θα φανεί παράδοξο τη στιγμή για την οποία υπάρχουν αρνητικά σχόλια την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις σχόλες, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αναλάβουν δεσμεύσεις, να συμμετάσχουν, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο ποιοτικά μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ πρέπει να πω ότι στο Ευρωπαϊκό Βασίλειο, στη χώρα μου, που όπως ξέρετε σε λίγο θα κάνει δημοψήφισμα εάν θέλουμε να παραμείνουμε εντός ή εκτός, το 2014 υπήρχαν περισσότερες αναφορές από, παρά από την Πολωνία και την Γαλλία που είναι ε, όσον αφορά τον πληθυσμό ισότιμες χώρες. Για πολλούς λόγους και πολύπλοκους. Αλλά ένα στοιχείο το οποίο και θα είμαι σύντομη, το οποίο πρέπει να τονίσω είναι ότι οι αναφορές θεωρούνται ως σημείο κλειδί αυτής της ε, δημοκρατικής συμμετοχής. Υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα ήθελα να φέρω. Για ποιο λόγο υποβάλλουν αναφορές οι πολίτες μας θέλουν να ακουστεί η φωνή τους. Πρώτα απ' όλα, είναι καλός τρόπος να ακουστεί η φωνή της. Μου είπε κάποιος αναφέρον ότι έτσι έχουμε την ε, δυνατότητα να μας ακούσει απευθείας ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ίσως το, το, ο χώρος στον οποίο καταβε, κατα, κατα, Φάνει ε, ο πολίτης στενοχωρημένος, είναι το ίστατο μέσο το οποίο διαθέτει, απογοητευμένος και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, διότι έτσι αισθάνονται οι πολίτες ότι τους ε, σεβόμαστε. Επίσης, πρέπει να πω ότι για τα ε, δικαιώματα των εργαζομένων οι αναφορές είναι πολύ καλές και για τα δικαιώματα απεργίας ή όχι. Πρέπει να πω όμως ότι όλο και περισσότερες αναφορές αναφέρονται στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Και έχουμε μιλήσει εδώ για τη σχέση μεταξύ χάρτου θεμελιωδών δικαιωμάτων και αναφορών που λαμβάνουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, μαζί με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ανθρώπων, διότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να ε, αυξήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών μας και τελικά να τους σταματήσουμε απόλυτα σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Το δικαίωμα αναφοράς νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει όλη αυτή τη διαδικασία το να ακούμε τους αναφέροντες να την ενισχύσουμε. Θα πρέπει πάντα η Επιτροπή να κάνει κάτι ε, με γρήγορο τρόπο, διότι πολλές φορές ε, χρειάζεται να περιμένουν οι άνθρωποι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πρέπει εφόσον πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο θεωρείται ως ένα θεμελιώδης δικαίωμα να επιταχύνουμε τις ε, διαδικασίες. Επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερη και στενότερη σχέση με τις εθνικές επιτροπές αναφορών που υπάρχουν σε διάφορες βουλές όπως το Κοινοβούλιο της Σκοτίας Φερυπής ή σε άλλες εθνικές συνελεύσεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε επίσης την σχέση που έχουμε με τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή και θα πρέπει όλοι οι ευρωβουλευτές από όπου και να προέρχονται να αναγνωρίσουν το ρόλο μας, να ε, είναι μαζί μας και να μας επιτρέψουν να φέρουμε με θετικό τρόπο και γρήγορο σε πέρας τις, ε, ε, τα καθήκοντά μας. Ευχαριστώ. Thank you very much παρέμβασή σας και θα ήθελα να καλωσορίσω στο σημείο αυτό την κυρία Μπεάτε Γκμίντερ, εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Έχετε το λόγο. Για πέντε λεπτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαστε εδώ σήμερα στην ακροασία αυτή να ανταποδώσω και εγώ τα, τους που ακούσαμε από την Επιτροπή σας προς τον διαμεσολαβητή. Να σας πω ότι είναι κάπως διαφορετικό φυσικά το πεδίο της εντολής μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα πρότυπα καλής διαχείρισης και χρηστής διαχείρισης μεταξύ όλων των ε, θεσμικών οργάνων, των σωμάτων και των ε, εξωτερικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχουν προβλήματα του κόσμου με την διοικητική πλευρά. Λαμβάνουμε καταγγελίες από πολίτες, εταιρείε ΜΚΟ, ενώσεις ε, εταιρικέ. Οποιοςδήποτε έχει δυνατότητα υποβολής καταγγελίας προς τον διαμεσολαβητή. 4.000 καταγγελίες λαμβάνουμε ένα έτος περίπου. Πολλές εξ αυτών, όπως και στην Επιτροπή Αναφορών, ε, δεν ταιριάζουν στο πεδίο των καθηκόντων μας και έτσι μας τιμώνει συχνά ο κόσμος, αλλά δεν έχουμε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αρμοδιότητα. Πρόκειται για πολιτική εφαρμογή, για παράδειγμα, της νομοθεσία, στα κράτη-μέλη ή για εγχώριες εθνικές πολιτικές και σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Οι 400 όμως βασικές καταγγελίες οι οποίες είναι παραδεκτές και όπου πραγματικά κάνουμε έρευνα, αυτές σε μεγάλη πλειονότητα έχουν να κάνουν με την έλλειψη διαφάνειας, με διαφάνεια, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη πρόσβασης σε έγγραφα, έλλειψη πρόσβασης και συμμετοχής. Σε πληροφορίες, πρακτικά, συναντήσεων και το καθεξής. Και αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους μας, να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε τη διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαμεσολαβητής ε, θέλει διαφάνεια σε όλες τις πολιτικές συναλλαγές για να βελτιωθεί και η ενημέρωση του πολίτη, γιατί μόνο όταν ξέρει κανείς τι γίνεται μπορεί να συμμετέχει καλύτερα και να κάνει τη φωνή του να ακουστεί στον πολιτικό διάλογο. Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που ερευνήσαμε είναι η έρευνα για το πώς οι σύναντες για την λήψη αποφάσεων ε, διαμορφώνουν τη διαφάνεια, που κατά πόσο είναι διαφανής σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, των τριμερείς διαλόγου του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου που συχνά διοργανώνονται με αποτελεσματικό τρόπο μεν, αλλά χωρίς την απαραίτητη διαφάνεια. Θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν η διαφάνεια και να κοινοποιήσουμε πιο πολλά στοιχεία με τους ενδιαφερόμενους. Είναι λοιπόν σημαντικό για μας να εισακούμε τις ανάγκες των πολιτών. Και αν δούμε τις, τις πολλές καταγγελίες που ακούμε, σημαντικό είναι να είμαστε, ε, να τους εισακούμε. Και νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε κακοδιαχείριση, αλλά συχνά ακούσαμε ε, διάφορα τέτοια παράπονα, διάφορες τέτοιες ενστάσεις και μας βοηθήσε αυτό. Είμαστε λοιπόν πολύ θετικοί για την επίλυση πολλών καταγγελιών που φτάνουν στο δικό μας επίπεδο και προσπαθούμε να προωθήσουμε περαιτέρω βελτίωση της διοίκησης έγινε και η στρατηγική έρευνα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και πιστεύουμε για παράδειγμα ότι θα έπρεπε να τεκμηριώσουμε καλύτερα να τεκμηριώνεται καλύτερα γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί για παράδειγμα μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο προτείνει μια συμβουλευτική ομάδα εργασίας και σε ό,τι φορά την συλλογή των ε, υπογραφών και επίσης εξετάζουμε τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο θέμα είχε να κάνει με τη διαφάνεια των διαδικασιών, των ε, συνομιλίων και την πραγματεύσεων για το TTIP, όπω ξέρετε. Για μας λοιπόν, βασικό σημείο εστίασης είναι η διαφάνεια, η συμμετοχή με τους πολίτες στις δικασίες αυτές και φυσικά θέλω να πω ότι με χαρά θα δεχόμασταν πιο πολλές καταγγελίες αν έτσι βοηθάμε τον κόσμο να βελτιώσει τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και την ποιότητα του Ευρωπαϊκού Διαλόγου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χμίντερ για την ε, παρουσία σας Τώρα, ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Καρλ Χάιντς Λάμπερτς, ο οποίος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. Καλώς ορίσατε κύριε Λάμπερτς και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν υπάρχει διάλογος θα πρέπει κάποιος να ομιλεί και κάποιος να ακούει. Και κατά προτεραιότητα θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες συμμετοχής εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη σήμερα διαπιστώνεται ότι βρισκόμεθα εις μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε Μιλάμε πολύ, αλλά δεν συνεννοούμαστε υπάρχει κάτι πάρα πολύ απογοητευτικό προς το παρόν και μετά από μισό αιώνα στην ε, Περιφερειά μου και στην Επιτροπή των Περιφερειών κατάλαβα το ότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι κάτι το πάρα πολύ ευάλωτο και τούτο διότι δεν έχουμε τις ίδιες αξίες. Να επομένως και θα πει διάλογος με τους πολίτες κάτι το οποίο με καίει γιατί εγώ προέρχομαι από την γερμανόφωνη κοινότητα του, ε, του Βελγίου εκεί στα σύνορα με τις κάτω χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία όπου την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης είναι κάτι για μας το καθημερινό και πρόκειται για ένα σοκ πριν από λίγους μήνες ξέρετε όταν είδα και πάλι να έχουμε ελέγχου στα σύνορα όταν πήγα να περάσω γιατί η τελευταία φορά που ε, θυμάμαι ήταν, ε, στη Γαλλία όταν ήμουν πάρα πάρα πολύ νέος. Οπότε θα πρέπει να διαπιστώσουμε την ανάγκη του να εμπλακούν και πάλι στην πραγματική οι Έλληνες πολίτες και θα πρέπει να στείλουμε και το μήνυμα. Για την Ευρώπη ποιοι μιλάνε περισσότερο σήμερα αυτοί που την αμφισβητούν. Είδατε τι έγινε στα τρία ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Είδατε σε ποιο σημείο ε, η Ευρώπη έχει γίνει για τους νέους ένας ε, εχθρός. Δεν είναι θέμα πια ε, μιας καλύτερης ζωής. Η Ευρώπη έχει γίνει κάτι που φοβίζει, γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει κάτι καινούργιο αφήγημα θα πρέπει επομένω να αλλάξουμε την ιστορική πορεία. Οπότε εδώ έρχεται ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών. Νομίζω μπορεί να τον ιδενοματίσει αυτό τον ρόλο, γιατί αναμφίβολα οι τοπικές και περιφερειακές αρχές από πολύ καιρό είναι ε, η πηγή της ε, συμμετοχής και η οργάνωση της συμμετοχής γίνεται όσο δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Οπότε γι' αυτό και πιστεύω ότι στη σημερινή κρίση το μήνυμα της Ευρώπης δεν πρόκειται να φτάσει στους νέους και δεν θα δουν θετικά την Ευρώπη Δεν θα απευθυνθούν στην Ευρώπη παρά μόνο εάν η συνάντηση γίνει σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Εκεί είναι πιο απλό, πιο προφανές κανείς να έρθει σε επαφή με τον δήμαρχό του πολύ πιο εύκολα από τον πρόεδρο τη Επιτροπής ή του Συμβουλίου, όσο και αν αυτή είναι υπέρ της άμεσης επαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βοηθάει το διάλογο με πολλούς τρόπους, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες επικοινωνίας και διαλόγου. Σήμερα δεν μιλήσαμε για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να αναφερθούμε επίσης σε όλες αυτές τις επαφές στα πλαίσια των προγραμμάτων όπως η Ευρώπη για τους ε, πολίτες, Ευρώπη για του πολίτη κλπ. Μιλάμε για δεκάδες και χιλιάδες προγραμμάτων που τα τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλα αυτά δεν αρκούν, άρα θα πρέπει να βρεθεί κάτι καινούριο, ούτως ώστε να είναι πιο ενεργός ο πολίτης και πιο συμμετοχή η δημοκρατία. Η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε ένα ψήφισμα που αφορά την επικοινωνία στο τοπικό επίπεδο που λέγεται να συνδέσουμε την Ευρώπη για με τους Ευρωπαίους και επομένως ε, θα πρέπει σε συγκεκριμένο πλαίσιο να πέθουμε στον κόσμο για την Ευρώπη με τρόπο που θα τους είναι κατανοητός για συγκεκριμένες καταστάσεις. Ε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Έχουμε ε, οργανώσει επομένως στο Ναμύρ, στο Βέλγιο, κάποιες εκδηλώσεις, στο στο Μιλάνο, ε, στη, στο σανανέρι της Ισπανίας, στο Βίλνιους της Λιθουανίας και πρόκειται για ε, κάποια συμπόσια συζήτηση, τοπικά και περιφερειακά και είδαμε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιεί τη, γλώσσα του πολίτη και όχι ε, την γλώσσα των τεχνοκρατών. κρατών. Ε, που να ακούτε τις συνεδριάσεις μας φεύγει πιο αποδομένος από όσο ήρθε. Άρα θα πρέπει έτσι να δείξουμε εμπιστοσύνη στον κόσμο. Και έτσι θα πιστέψουν στην προσθέμενη αξία της Ευρώπης. Το μάλλον κατά όλες οι σημερινές ε, προκλήσεις όπως το προσφυγικό, όπως η ενεργεια των νέων, όπως ε, το, το, το, το γκρέμισμα της Ευρώπης μέσα από το Brexit και από άλλες απόπειρες γκρεμίσματος ε, θα αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από μια κουλτούρα, ένα πνεύμα συμμετοχής. Είναι ένα εργαλείο για να βελτιώσουμε την ε, νομιμότητα, την νομιμοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων. Άρα εδώ θα μπορούσε να πει κανείς πολλά. Και κυρίως δεν θα πρέπει βέβαια κανείς να απογοητεύεται. Πάρα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι βέβαια στην ηλικία μου δύσκολο να αλλάξω αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο άλλη εναλλακτική. Μόνο η ευρωπαϊκή οικοδόμηση και κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να επιληθεί από μια χώρα από μόνη της όσο μεγάλη και αν είναι αυτή ή ακόμα και αν είναι μικρή δεν λέει τίποτα αυτό. Άρα θα πρέπει να πλησιάσουμε τον κόσμο και άλλα είπαμε να πολλαπλασιάσουμε στην Επιτροπή Περιφερειών τις προσπάθειές μας για αυτό τον σκοπό και ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το πνεύμα συμμετοχής, θα πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ε, με εκδηλώσει όπως κάναμε στην Αστούρια ή όπως είπαμε στη Βαλονία και έτσι να πάμε για καινούργιες μορφές συμμετοχής. Ξέρω ότι πρόκειται για μια μάχη, ακόμα δεν έχουμε κερδίσει, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στην Ευρώπη την ε, θέση που της ε, αρμόζει ούτως ώστε να μπορέσει να λύσει τα σημερινά αλλά και τα αυριανά προβλήματα. Κύριε Λάμπερτ, σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα δώστε το λόγο στον κύριο Ζων Πολ Γκοζές, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ρόμπερτ Σούμαν. Σωστά τα είπα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε. Έχετε το λόγο, λοιπόν. Δεν θα επανέλθω στους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Η θέση σε εφαρμογή είναι κάτι το οποίο ήδη έχει λεχθεί τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία προσπαθεί να βρει μέσα για να εκφράσει καλύτερα τις προσδοκίες των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία είναι μέσον εκδημοκρατισμού και δυναμισμού των ε, αποφάσεων που λαμβάνονται στην Ευρώπη. Για να έχει θετικά αποτελέσματα και να τα αισθανθεί ο πολίτης είναι απαραίτητο να κάνουμε παιδαγωγική δουλειά. Έχουμε παιδαγωγικό έργο να φέρουμε σε πέρας προς τους πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αυτή την περίοδο που όπως υπενθυμίστηκε είναι περίοδος που ε, έχει πολλά σκαπανεβάσματα η ιδέα της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό σχέδιο πιο απαραίτητο από ποτέ θα πρέπει πραγματικά να έχει μια νέα όφηση η οποία δεν θα μπορέσει να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες παρά μόνον θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι εάν διαδίδονται πληροφορίες σε τακτά διατήματα για το τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη. Εάν δείξουμε με επιχειρήματα τι ακριβώς κάνουμε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτούς που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις και εάν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ποιοτικά στις προ... Στε να δώσουμε απαντήσει στι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι πρωτοβουλίε όλων αυτών που θέλουν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιδέα και να δεστοποιήσουμε τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και με ανταποκριτές σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, το Ίδρυμα Σούμαν αναγνωρίζεται ως μία εγκεκριμένη φωνή όσον αφορά την ιδέα της Ευρώπης. Έχει φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της ε, από τότε που ιδρύθηκε με διαφάνεια και με συνεχή τρόπο. Αλλά ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση του Ιδρύματό μας είναι όλο και πιο δύσκολη. Πολλά σχέδια και μελέτες για την πολιτική μετανάστευση που αφορούν τους πρόσφυγες ή ακόμη τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων τις ιδρύματά μας. Για το λόγο αυτό το Ίδρυμά μας καθώς και όπως άλλα ε, ιδρύματα όπως το Ινστιτούτο Ζακ Τελόρ πρέπει να επωφεληθούν από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε τοπικό επίπεδο αυτό το παιδαγωγικό ρόλο στη Γαλλία έχουν αναλάβει τα σπίτια της Ευρώπης που είναι μέλος μιας συνομοσπονδίας και από το δίκτυο η Ευρώπη απευθείας. Πρόκειται για οργανώσεις που πραγματικά και εκείνες δεν έχουν τα μέσα που τους χρειάζονται και ε, παίρνουν τους πόρους που χρειάζονται από τις δημόσιους πόρους που βρίσκονται σε μείωση. Εξάλλου πρέπει να πω ότι είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι πολίτες και από τα πολιτικά κόμματα. Ελέγχθη αυτό προηγουμένως και δεν θα επανέλθω. Δεξιά και αριστερά η Ευρώπη πολλές φορές λαμβάνεται μόνο υπόψη από τα ε, κόμματα πολιτικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιεί από αποδιοπομπαίος τράγο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Εξάλλου τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως και στις περισσότερες γαλλικές χώρες ε, με πολύ, ε, σε πολύ μικρό ποσοστό αναφέρονται στην Ευρώπη. Πρόσφατα οι βουλευτές Καρές και της ε, Γαλλικής Συνέλευσης είπαν ότι θα πρέπει τα διάφορα θέματα με τα οποία ασχολείται η Ευρώπη να αποκωδικοποιηθούν για να τα καταλάβουν καλύτερα όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν συμπληρωματικές προσπάθειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκόζες. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Άσια Καβράκοβα, Διευθύντρια της ε, Υπηρεσίας ΙΚΑΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράσης των Πολιτών. Έχετε το λόγο κυρία Καβράκοβα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όλη μέρα σκέφτομαι. Τι γίνεται όσον αφορά αυτό το οποίο λέμε αν είναι καλό ή κακό για την πρωτοβουλία, γιατί είπαμε ότι από το πρωί αυτά τα οποία ακούμε, νομίζω ότι είναι κάτι το θετικό, γιατί η αποστολή του φορέα μας είναι οι άνθρωποι και οι πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Επί 25 χρόνια έχουμε στρατευτεί σε αυτόν τον σκοπό και έχω να σας πω τα εξής τρία. ή 3,5 θέματα. Έχουμε βασίσει στο Ευρωβαρόμετρο και λέει ότι 58% των Ευρωπαίων δεν έχουν ιδέα για το τι θα κάνουν σε περίπτωση που καταπατηθούν τα δικαιώματά τους. Η απάντηση είναι η εξής. Θα πρέπει να, να αναζητήσουν συμβουλή. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύστημα καταράκτη γιατί μόνο ένας μίλησε γι' αυτό το πρωί, την επίλυση του προβλήματος. Είπαμε ότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργούν τα εργαλεία που υπάρχουν. Δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ψάχνουμε για κάτι καινούργιο. Οπότε έχουμε το σύστημα αυτού του της πύλης και εκεί μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για κάθε δικαίωμα κάποιου Ευρωπαίοι. Αν αυτό δεν αρκεί για να λυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, τότε έχουμε την υπηρεσία μας. Europe Advice ονομάζεται. 19 χρόνια λειτουργεί και έχουμε συμβούλους νομικούς και αυτοί μπορούν να συμβουλεύσουν τους ε, Ευρωπαίους όποτε έχουν κάποιο πρόβλημα για κοινωνική πρόνοια, ε, δημόσια υγεία, ε, το να ιδρύσουν μια εταιρεία, σχέση με θεωρίες διαβατήριων, έχουμε 60 νομικούς συμβούλους. Είναι ένα δίκτυο σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτοί δωρεάν παρέχουν νομικές συμβουλές σε όλες τις ε, επίσημες γλώσσες των ε, κρατών μελών. Οπότε και έχουμε δώσει τις πληροφορίες σε 22.127 Ευρωπαίους, δηλαδή 9,5% αύξηση σε σχέση με το παρελθόν που βλέπουμε τα κράτη-μέλη. Ε, λένε και πιο πονηρά είναι όσον αφορά το πώς θα καταπίτουν αυτά τα δικαιώματα, αλλά και οι πολίτε χρειάζονται περισσότερε συμβουλέ, Υπάρχει υπηρεσία του συμβουλές και η επόμενη φάση αυτού του συστήματο Cascade, που το λέμε, προχωρεί, όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δημόσια διοίκηση. Και έχουμε επομένως αυτή τη διοικητική πύλη, ούτω ώστε να ερχόμαστε σε επαφή. Μία υπηρεσία που νομίζω είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, να τη μάθουν οι Ευρωπαίοι. Είδαμε μόνο στα αποτελεσματικά της ε, στατιστική που λέει ποια είναι τα βασικά δικαιώματα που τα αγνοούν. μεταξύ των οποίων και τα εκλογικά δικαιώματα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Όταν απαντούν οι νομικοί συμβούλοι μπορούμε να τους δίνουμε κάποιον σύνδεσμο και έτσι αυτοί τουλάχιστον 22.000 και τόση πολίτες που προσφεύγουν στην υπηρεσία μας να έχουν και αυτή την παραπάνω πληροφορία όσον αφορά αυτό το δικαίωμα, το εκλογικό. Να, στο φροντίσει η Γενική Διεθνή. Τώρα, ένα άλλο θέμα, ένα άλλο εργαλείο. Κατ' ανακάλυψα πρόσφατα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι γνωστό. Έτσι, εμπειρικά, για μου. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πλατφόρμα διαδικτυακή που ονομάζεται το, το, το, δίκτυο, το, διαδίκτυο ένα site που λέει ότι μπορούν οι πολίτες να δουν την νομοθεσία πώς μπορούν να βελτιώσουν την νομοθεσία πώς μπορούν να την προσαρμόσουν στις ανάγκες τους και να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Πόσοι από εσάς το γνωρίζετε, σηκώστε το χέρι σας. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Λέει ο πρόεδρο, Μην, μην, αντιδράτε. Όχι, όχι, δεν ήταν η ρητορική η ερώτηση, λέει η κυρία Κάβα. Εγώ θα πράγματα που πείτε γιατί δουλεύω πάνω σε αυτή την πλατφόρμα για την καλύτερη νομοθεσία. Και με αυτή την πλατφόρμα έχουμε λάβει 250 προτάσεις για καλύτερη νομοθεσία. 99% αυτών προέρχονται από επιχειρήσει. Γιατί αντίθετα οι πολίτες επιχειρήσεις τα ξέρουν αυτά. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμο. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει και για τους πολίτες και όχι μόνο μόνο για τις επιχειρήσεις να βελτιωθεί η νομοθεσία. γιατί βέβαια ενδιαφέρονται για αυτή την πλατφόρμα και οι εθνικές αρχές. Οπότε, κάντε τον κόπο, ρίξτε μια ματιά σε αυτή την πλατφόρμα και πέστε το στους γνωστούς σας. Τώρα έχουμε και το θέμα της διαβούλευσης γιατί είδα και ένα στιγμό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω 80% των Ευρωπαίων θεωρούν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία της συμμετοχής για τέτοιες διαβουλεύσεις, κυρίως οι ναι, νέοι. Συμφωνώ. Αλλά έχω να σας πω ότι όπως γίνονται οι διαβουλεύσεις από την Επιτροπή σήμερα, δεν εξυπηρετούν τους πολίτες παρά μόνο τα οργανωμένα συμφέροντα. Καλά μέχρι εδώ. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποια συμπληρωματική παράλληλη διαδικασία που να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ε, πολιτών και να εμπλέκονται επομένω. ας πούμε για τους νέους ε, και συμφωνώ με τους ανθρώπους από το Φόρουμ των Νέων είναι δεν απευθύνονται αυτοί στους λαμβάνοντες αποφάσεις το ανάποδο θα πρέπει να γίνεται θα πρέπει οι λαμβάνοντες αποφάσεις να πάνε να μιλήσουν στον κόσμο, στους νέους, να το κάνουν δηλαδή, είτε κυριολεκτικά είτε με κάποιο τεχνικό άλλο τρόπο. Έχουμε επίσης 25 ε, παραδείγματα sourcing Νομοθεσία για crowdsourcing. Καινούριο θέμα. Και αυτό αφορά μια πρωτοβουλία πολιτών. Και εγώ πιστεύω πως και άλλοι ότι θα πρέπει η σχετική νομοθεσία να αναθεωρηθεί τώρα και όχι αύριο. Και κάτι άλλο το οποίο το έχουμε παραλείψει αλλά έπρεπε να αναφερθεί, να αναθεωρήσουμε νομοθεσία ώστε να μπορούμε να έχουμε ε, περισσότερους που εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους. Αν τα κάνουμε αυτά νομίζω ότι πάμε για περισσότερη απογοήτευση. Ευχαριστούμε κύριε Καβρακόβα πολύ παιδαγωγικά αυτά τα οποία μας είπατε. Σας ευχαριστούμε. Ήταν η τελευταία από τα μέλη του πάνελ που έλαβαν το λόγο και σας ευχαριστούμε όλους για τα όσα μας είπατε που ήταν τόσο ενδιαφέροντα. Και τώρα, όποιος θέλει μπορεί να υποβαλεί ερωτήσει και να υπάρξουν απαντήσεις από το πάνελ. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι για να μπορέσουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερους έχει ο καθένας, μια που θα είναι τόσο γενναιόδωρα θα δώσω τρία λεπτά. Τρία λεπτά στον καθένα. Ρωτήστε ελεύθερα ερωτήσεις, πέστε τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας, αλλά όχι για παραπάνω από τρία λεπτά λέει ο πρόεδρος. Έχουμε κατάλογο αυτών που ζήτησαν το λόγο. Δεν βλέπω το όνομά σα, αγαπητή κυρία. Με εσεί πίσω-πίσω, ναι, είναι επειδή δεν έχω ταμπελάκι να συστηθώ. Άλεξ Ενδρίνα Ναμόβιτ από το European Civic Forum, ε, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πάνω από 100 ενώσεων στην Ευρώπη για την συμμετοχή των πολιτών για την προάσπιση του χώρου των πολιτών για να ακουστεί η φωνή των πολιτών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε την, ε, το θέμα αυτό των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά με προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τώρα που και τελειώνει η ημέρα δεν έχω ακούσει ούτε έναν να μιλάει για την οργάνωση των πολιτών στα οργανωμένα πολιτικά δικαιώματα και όντω. Αν παραμείνουμε στο πλαίσιο του άρθρου 20 και των δικαιωμάτων που συνδέονται με την κινητικότητα, όντω ε, έχουμε να κάνουμε με τα μεμονωμένα άτομα, με τους μεμονωμένους πολίτες. Αλλά νομίζω ότι στι ευρωπαϊκέ συνθήκε και ιδιαίτερα στη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουμε πάρα πολλέ άλλε ευκαιρίε και δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν με τα πολιτικά δικαιώματα. Ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατέστησε πρωτογενέ δίκαιο, το άρθρο 11, το οποίο όντω ε, σε ό,τι αφορά την μεμονωμένη συμμετοχή μέσω της πρωτοβουλία του πολίτη αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και με βέβαια το γνωρίζετε όλοι σας στο γεγονός τη συμμετοχή των οργανωμένων πολιτών μέσω οργανώσεων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στην υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να διεξαγάγουν ανεκτό και διαφανή διάλογο με τις ενώσεις αυτές. Εμείς επί χρόνια εργαζόμαστε ως οργάνωση και συλλογικά με πολλές άλλες οργανώσεις παρόμοια με τη δική μας. Κοιτώντας και πώς διοργανώνεται η συμμετοχή του πολίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάνουμε συστάσεις, αντιδρούμε και συμμετέχουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις και είμαστε μεταξύ των οργανώσεων εκείνων που έχουν διατυπώσει και συγκεκριμένε προτάσει. Ελπίζουμε πραγματικά αυτή τη φορά το όραμα αυτό του πολίτη να προβληθεί σε ό,τι αφορά τις ε, ενώσεις των πολιτών. Αν χρειαστεί, έχουμε και <coughs> συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό το έγγραφο που βλέπετε βάσει των εμπειριών μας μέσω του Ευρωπαϊκού του Εθελοντισμού, του Ευρωπαϊκού Ετου του Πολίτη και τον πολιτικό διάλογο με τι πολιτικέ ενώσει και τα πολιτικά κινήματα. Και κάποιοι από εσά, θα το γνωρίζετε άλλωστε. Δυστυχώ δεν είναι κανεί εδώ από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ελπίζω όμω να είναι κάποιοι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας μιλήσουν και να μας διαβεβαιώσουν ότι οι ανησυχίες αυτές οι οποίες εκφράζονται εδώ και χρόνια θα βρουν μια απάντηση στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ένας κύριος εκεί πίσω. Α, όχι, δεν θέλετε το λόγο. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Όλα είναι σαφή και ξεκάθαρα. Είσαστε εξαιρετικοί. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και για τις παρεμβάσεις σας. Και τώρα να ακούσουμε τα καταληκτικά σχόλια. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Τίνα Εστόλα, Γενική Διευθύντρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη Καταναλωτών και Ισότητα Φίλων. Η κυρία Αστόλα, λοιπόν, να έχετε το λόγο. Δεν σας έβλεπα. Άξιοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που μπορώ να κάνω τα καταληκτικά αυτά σχόλια, τα απορίσματα να διεξαγάγω για το πως μπορούμε να αναπτύξουμε στο έπακρον την ιδέα των ευρωπαϊκών πολιτικών δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντική και επίκαιρη η χρονική στιγμή συζήτηση μετά τις διαβουλεύσεις και μετά από αυτά που δημοσιεύτηκαν στο Ευρωβαρόμετρο. Και να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις κοινέ μας αξίες, να βελτιώσουμε περαιτέρω τη δημοκρατική συμμετοχή και να κάνουμε τη ζωή των ε, Ευρωπαίων πολιτών πιο εύκολη. Μας είπαν λοιπόν ότι θέλουν να ακουστούν οι πολίτες και ότι θα πρέπει να κάνουν πιο πολλά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, όντως χρειάζεται να προασπίσουμε τις κοινές μας αξίες, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την συμμετοχή, την διαφορετικότητα και το καθεξής. 90% πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνει πιο πολλά για να προωθηθούν οι κοινές αξίες στο σχολείο, μεταξύ της νεολαίας, στην κοινωνία, στο σύνολό τη. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων των κρατών μελών, δηλαδή, αλλά και των τοπικών περιφερειακών αρχών. αλλά ασφαλώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό ζητούν οι πολίτε αυτό ζήτησαν και στι διαβουλεύσει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον την ευρωπαϊκή αυτή ηθαγένεια. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, ξέρουν σήμερα πιο πολλά για την ευρωπαϊκή αυτή ηθαγένεια παρά ποτέ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αρκεστούμε σε αυτό και όπως είπε και η Επίτροπος Γιούροβα το πρωί στα εισαγωγικά σχόλια, η ηθογένεια δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό οικοδόμημα. Όχι, δίνει και στους πολίτες συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Το να είναι κανείς Ευρωπαίος πολίτης θα έπρεπε να συνεπάγεται ότι αισθάνεται στο σπίτι του σε οποιοδήποτε μέρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναλάβουμε πιο συγκεκριμένε δράσει για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Συχνά οι πολίτε, βλέπετε, δεν συνειδητοποιούν απόλυτα τα δικαιώματά του και αυτό το ακούσαμε και στην ε, αμέσω προηγούμενη παρέμβαση και ω πολίτε δεν γνωρίζουν απαραίτητα τι θα πρέπει να κάνουν όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του, Αντιμετωπίζουν δυσκολίε όταν ασκούν τα δικαιώματά τους στην πράξη και συχνά οι δυσκολίες αυτές έχουν να κάνουν με μακροχρόνιες και βαριές διαδικασίες έλλειψη πληροφορίες και το καθεξής. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορεί να διευκολυνθεί η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Α, από ό,τι κατάλαβα, έχουν συζητηθεί εδώ σήμερα πολλές ε, καλές ιδέε, για παράδειγμα πληροφόρηση και βοήθεια για την απάντηση στις ερωτήσεις που προκύπτουν όταν κάποιο εγκαταστάται σε μια καινούργια χώρα και το πώ να καταχωριστεί κτλ. Η ελεύθερη μετακίνηση αποτελεί μια ευκαιρία για τους πολίτες που ταξιδεύουν, δουλεύουν, σπουδάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή γνώμη καταδεικνύει ότι οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα στατικό αντίκτυπο και για την πρόοδο και για την ανάπτυξη και για την οικονομική ανάπτυξη. 71% πιστεύουν ότι η ελεύθερη μετακίνηση έχει οικονομικά ωφέλη για τη χώρα τους. Και η ελεύθερη μετακίνηση αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δικαίωμα το οποίο εκτιμούν οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει λοιπόν το δικαίωμα αυτό να λειτουργεί ακόμα καλύτερα για το προς των πολιτών και της απασχόλησης και αντιμετωπίσει ό,τι τυχόν προβλήματα παραμένουν και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τους κανόνες και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την ανταλλαγή των πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια με τους νέους κανόνες για την νέα κυκλοφορία α, και της προξενικής προστασίας. Αυτό αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για να εφαρμοστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα αυτό. Προστασία δηλαδή σε τρίτες χώρες όταν ο πολίτης ε, τη χρειάζεται. Όπως καταδεικνύεται και από το Ευρωβαρόμετρο, αυτά τα προξενικά δικαιώματα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό ή πολύ κατανοητό από τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε λοιπόν περιθώριο πολύ μεγάλης περαιτέρω επεξήγησης της νέας αυτής νομοθεσίας. Κυρίε και κύριοι, να πω και δύο λόγια για τα πολιτικά δικαιώματα όπως προκύπτει και από την έκταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 για τις ευρωεκλογέ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, προσπάθειές μας και να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογέ και θα πρέπει αυτό να έχει στο στόχο στο βασικά τους νέους. Και όπως είπε και η Επιτροπή το πρωί, θα πρέπει αυτό να ξεκινήσει τώρα. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, χρειαζόμαστε καλύτερη πληροφόρηση για το ποιε ε, είναι οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και τι συνέπεια έχουν για την καθημερινή ζωή των πολιτών. Οι πολίτε το έχουν ζητήσει αυτό. Θα πρέπει να ε, ευαισθητοποιήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη για τα δικαιώματά του και αν πετύχουμε αυτό θα πετύχουμε και πιο ενεργή δέσμευση των πολιτών σε ό,τι αφορά και τις εκλογές του 2019 η πολιτική νομιμοποίηση σε ό,τι αφορά τους κορυφαίους υποψηφίους, τους πίθεν καντιντάτ, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα και η μεταρρύθμιση του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου, του νόμου για τις εκλογές του 72 αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Είναι επίσης σημαντικό να καταστεί πιο απλό να συμμεταχεί κανείς στις ευρωεκλογέ και στις τοπικές εκλογές. Οκτώ στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι θα ήταν πιο απλό να ψηφίσουν αν ακολουθούνταν κάποιες καλές πρακτικές παντού. Και θα πρέπει λοιπόν να προωθηθούν επιτέλους αυτές οι βέλτιστες οι οποίες ήδη εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων για τις καρποφόρες συζητήσεις που διεξήχθησαν σήμερα και για τις νέες ιδέες που παρουσιάστηκαν προκειμένου να μεταφραστούν οι ιδέες των πολιτών σε πρακτικά μέτρα. Θα επεκτείνουμε λοιπόν θα τις διευρύνουμε τις συνδέσεις αυτές και θα καταθέσουμε φέτος ήδη συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένες βάσεις στην επόμενη έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγέννηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το σημερινό σας έργο. Και πολύ λυπάμαι που δεν ε, ήμουν εδώ όλη την ημέρα. Ευχαριστούμε κύριε Στόλα για την παρέμβασή σας, που δεν είναι τελική. Κάνατε κάποιες ε, ε παρατηρήσεις τελειώνοντας τη μέρα, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο για το διατάφτα στην ε, πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών την κυρία Βαλξον. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σα λόγια. Όπω αρχίσαμε σήμερα το πρωί, έτσι και τελειώνουμε. Αγαπητά μέλη, ομιλητές, συμμετέχοντε, με ευχαρίστηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σας πω ότι οργανώσαμε αυτή την ακρόαση στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτρόπου σα, του ε, συνοδεργανωτές, του συναδέλφου από τις τρει άλλες κοινοβουλευτικέ επιτροπές για να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους, τους εμπειρογνώμονες, τους αναφέροντες που πραγματικά συνεισέφεραν θετικότητα στις σημερινές συζητήσεις. Ελπίζω ότι τώρα όλοι αισθανόμαστε αρκετή έμπνευση μετά από αυτά που διεμήφθησαν και με κουράγιο θα προσπαθήσουμε περαιτέρω να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα. Χαίρομαι διότι οι συνάδελφοι που δεν είναι μέλη της Επιτροπής Αναφορών αλλά μέλη άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών είχαν σήμερα το προνόμιο να ακούσουν κάποιους από τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ και να μας εκθέσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα και τένιες οι συνεισφορές τους είναι πραγματικά μεγάλη πηγή ενημέρωσης για μας που είμαστε οι συνομοθέτες σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι με την εξαιρετική μας γραμματεία και με τους υπεύθυνους των τμήματων θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών και να αναφορέσουμε τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κάποιοι ανέφεραν σήμερα και ε, παραθέτω, τι κάνουμε σήμερα. Ασχολούμαστε με το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα. Εξαιρετική έκφραση. Πολλές φορές λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε δικαιώματα και ως καταναλωτές στην Ευρώπη και εμείς ως πολιτικοί εκλεγμένοι στην Ευρώπη κοιτούμε πολλές φορές τους πολίτες μόνο ως ψηφοφόρους. Ας το σταματήσουμε αυτό. Όλοι είμαστε πολίτες. Οι εκλεγμένοι, οι καταναλωτές, όλοι μας κάποιες φορές και επίσης κάποιες φορές αναφέροντες. Όλοι όμως είμαστε πολίτες και εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλούμε για ψηφοφόρους και να απευθυνόμαστε διαφορετικά στους συμπολίτε μας, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον ο διάλογος μεταξύ μας. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται σε θέματα ηθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη. Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες τον διάλογο μεταξύ μας. Ακόμη και πάλι θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους για τη συμμετοχή σας, για την ε, παρουσία σας και μην διστάζετε να απευθύνεστε σε εμά όταν έχετε ένα θέμα το οποίο πρέπει να θέσετε υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γεια σας, καλό βράδυ.